Εγώ λοιπόν καλωσορίζω όλους και όλες τις συμμετέχουσες εδώ σε αυτή την ε, ακρόαση, δημόσια ακρόαση για θέμα για το πώς η φτώχεια πλήττει τις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν κυρίως να στραφώ προς την, την κυρία Φράμ που είναι αρμόδια εισηγήτρια και τις εμπειρογνώμονες που καλέσαμε εδώ. Επίσης να καλωσορίσω εκπροσώπηση από την Επιτροπή που έχουμε εδώ στη συνεδρίασή μας. Επίσης να πω ότι έχουμε και μια ομάδα επισκεπτών από την κυρία Πλάμ που συμμετέχουν σήμερα. Καλωσορίζουμε λοιπόν και τους επισκέπτες για αυτήν εδώ την ακρόαση και να πω ότι ελπίζω να έχουμε ένα σωστό, επικοδομητικό διάλογο για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Άλλη μια φορά λοιπόν σας καλωσορίζω και ελπίζω όλοι να έχουν στα χέρια τους αυτά εδώ τα έγγραφα που κρατώ στα χέρια μου που ε, είναι ένα σύνολο σελίδων που αφορούν το σημερινό θέμα και ελπίζουμε όλες και όλοι να το έχουν λάβει. Έχουμε λοιπόν το έχουμε το πρόγραμμα ως εξή. Θα υπάρχουν δύο πανέλ συζητήσεων. Το πρώτο που έχει να κάνει με τις διαστάσεις της φτώχειας και τις επιπτώσεις στις γυναίκες. Αυτό είναι το πρώτο μέρος της ακρόασης που θα έχουμε. Στο δεύτερο μέρος έχουμε ένα άλλο θέμα, δηλαδή τον γενικότερο τον ε, στόχο μας για να μειώσουμε την φτώχεια και ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μαζί όμως σήμερα και είναι σημαντικά θέματα. Όλοι και όλες ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή ζούμε μια κατάσταση όπου η, η φτώχεια πλήττει περισσότερο τις γυναίκες και γι' αυτό αποτελεί ένα από τα θέματα που είναι προτεραιότητα για μας και δεί για τη σημερινή ακρόαση και η κυρία Πλάμ, όπως ξέρουμε, έχει ανα... είναι υπεύθυνη για μια έκθεση πρωτοβουλίας με αυτό εδώ το θέμα. Με αυτά λοιπόν ε, εύχομαι να έχουμε μια σωστή επικοδομητική συζήτηση και αμέσως θα δώσω το λόγο στην κυρία Πλάμ για να κάνει κάποια σχόλια ε, σαν εισήγηση θα έλεγα. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Thank you, Chair. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους. Τιμή μου, μεγάλη μου τιμή που είμαι συγγήτρια πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό. Θα ήθελα να ευχηθώ ένα θερμός καλώς ήρθατε στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στους εμπειρογνώμονες, σε όλους τους φιλοξενούμενους μας και χαιρετίζω και τους συναδέλφους μου και ιδιαίτερα τους αγαπητούς φίλους από τη Ρουμανία, από το Σοσιαλδημοκρατικό από την οργάνωση γυναικών του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της χώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χρησιμοποιήσω τώρα τη μητρική μου γλώσσα, αν μου επιτρέπετε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα εν ώψη της ε, κατάστασης που επικρατεί στην Ευρώπη σήμερα και που προκλήθηκε κυρίως από την ε, οικονομική κρίση, τη χρηματοπιστωτική κρίση και που επιβαρύνει ιδιαίτερα στις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για την επεξεργασία αυτής της έκθεσης και θα μας ε, δώσει την δυνατότητα να συμπεριληφθούν οι εμπειρίες αυτές που σχετίζονται με το φαινόμενο της φτώχειας, της θέσης φτώχης όπως πλήττει τις γυναίκες στην Ευρώπη και επίσης τις βέλτιες ε, πρακτικές που είναι αναγκαίες ώστε να περιοριστεί η φτώχεια. Ενώπιση του γεγονότο ότι το έτο 2010 είναι το ευρωπαϊκό Έτο για την καταπολέμηση τη στόχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού, θα πρέπει να επιστήσουμε την ε, προσοχή μας στις ε, γυναίκες ανεξάρτητα από το κατά πόσο πρόκειται για γυναίκες στο πλαίσιο μιας μονογονεϊκής οικογένειας ή γυναίκες που επιστούν μια θέση εργασίας ή είναι μετανάστριες. Σήμερα οι γυναίκες πολύ συχνά βρίσκονται σε καταστάσεις με υψηλό κίνδυνο φτώχειας. Όταν είναι έγκυες, για παράδειγμα, δεν έχουν την δυνατότητα πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή επειδή έχουν ε, δουλέψει όλη τους τη ζωή μόνο στο σπίτι, μια δραστηριότητα η οποία δεν αμείβεται και η οποία τελικά οδηγεί σε συρρήκνωση των οικονομικών πόρων. Και υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτή την κατάσταση και βάσει των στατιστικών στοιχείων ο κίνδυνος της ε, φτώχειας για γυναίκες που να φρέφουν μόνες του τα παιδιά τα παιδιά τους είναι τριπλάσιος από τις γυναίκες που ζουν σε κανονικές οικογένειες. Και η κατάσταση αυτών των, γονεϊκών, ε, των γυναικών συγγνώμη, είναι συχνά πολύ πιο δύσκολη, δύσκολη από ό,τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία. Σε σχέση με τους άνδρες, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολύ ψηλότερο κίνδυνο αποκλεισμού, κοινωνικού αποκλεισμού από τους άνδρες. Και αυτό ισχύει κυρίως για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας για τις οποίες το 2008 ο κίνδυνος αυτός αυξήθηκε, κατά, αυξήθηκε στο 22% σε σύγκριση με το 16% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό για τον ανδρικό πληθυσμό. Και αυτό το ποσοστό αυξάνεται στο 35% για γυναίκες ε, που είναι μετανάστριες. Υπάρχουν μια σειρά από κοινωνικούς ε, δείκτες οι οποίοι επισημαίνουν αυτά τα φαινόμενα και ο δικός μας ρόλος είναι να ε, παροτρύνουμε τους πολιτικούς να λάβουν κάποια μέτρα. Πέραν τούτου, οι ενέργειες οι οποίες έγιναν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των προσπαθειών μας για να μπορέσουμε να δώσουμε μια έμφαση στο φαινόμενο της στόχιας. Αλλά βέβαια θα πρέπει να συγκεντρωθούμε σε ειδικά μέτρα, ιδιαίτερως εκείνα τα μέτρα που εξασφαλίζουν για τις γυναίκες μια ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας και επίσης την ε, προσπάθεια μείωσης της ε, φτώχειας μεταξύ των ε, γυναικών. Επίσης θα πρέπει να συγκεντρωθούμε σε μέσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ε, στρατηγικές που συμπεριλαμβάνουν τη διάσταση της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων και που θα πρέπει να συμπεριφθούν σε όλες τις ε, πολιτικές που χαράσουμε. Δεν θα πρέπει να παραμελούμε τις επιπτώσεις της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού γιατί όλα αυτά καθιστούν τις γυναίκες μια αδύναμη κατηγορία του πληθυσμού που πολύ συχνά πέφτει θύμα εμπορίας ε, ανθρώπων ή βίας. Και ε, η πραγματική κατάσταση δυστυχώ δεν ε, εκφράζεται μέσα των στατιστικών στοιχείων. Και τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σήμερα δεν στοχεύουν στην ίση μεταχείριση των δύο φύλων και δεν είναι προσαρμοσμένα στην ιδιαίτερη κατάσταση του γυναικείου πληθυσμού. Η σταδιακή παρουσιάζουμε μας δίνει τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουμε τις πραγματικές διαστάσεις της φτώχειας και να τις συμπεριλάβουμε στις πολιτικές μας και επίσης μας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις αυτής της κατάστασης οι δικές σας εισφορές, οι δικές τοποθέτησεις έναντι των ισχυουσών πρακτικών και πολιτικών είναι σημαντικές σε σχέση με το τρόπο που διαμορφώνεται, για παράδειγμα, η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και επίσης σε σχέση με τα θεσμικά όργανα τα οποία θα πρέπει μελλοντικά να συμπεριληφθούν για την επεξεργασία αυτής της στρατηγικής. Και όλα αυτά θα μας καταδείξουν τα προσεχή βήματα τα οποία θα πρέπει να κάνουμε στο πλαίσιο αυτών των στρατηγικών. Έναψη της ανακοίνωσης στρατηγικής όσον αφορά τη στρατηγική της Ένωσης για το 2020 αναφέρονται οι στόχοι. Μεταξύ αυτών είναι η μείωση των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από το αέριο της φτώχειας κατά 20%. Αυτό σημαίνει 20 εκατομμύρια άνθρωποι λιγότεροι θα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας εφόσον επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Και το μέτρο αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε πολιτικές που έχουν σαν στόχο την προστασία των γυναικών από την φτώχεια. Είμαι απολύτως πεπισμένη ότι ο ρόλος αυτής της ακρόασης θα είναι ακριβώς ε, αυτός, δηλαδή να μας δώσει ένα προσανατολισμό ούτω ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση των γυναικών που ζουν μέσα στη φτώχεια και να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα για να εκπληρώσουμε αυτόν τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή την κρόαση. Είμαι πεπισμένη ότι όλες οι απόψεις που θα ακουστούν εδώ από συναδέλφους και από εμπειρογνώμονες θα συμπεριληφθούν σε μια έκθεση πρωτοβουλίας. Και θα ήθελα κυρία Πρόεδρε να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Eh, Ευχαριστούμε την κυρία Πλάμπ.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 Λοιπόν, ας ξαναρχίσουμε. Ε, και ελπίζω όντως η διερμηνία να λειτουργήσει. Λυπάμαι ειλικρινά που είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα και περιμέναμε, αλλά ήταν καθαρά τεχνικό. Τώρα ας ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχει συνέχεια και να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας στις διαφορετικές μητρικές μας γλώσσες. Λοιπόν, καλωσορίζω την κυρία Ρεγίνα Βουέμπχοφερ, η οποία είναι συντονίστρια στο Women Against Violence in Europe. Παρακαλώ, κυρία Βουεμπχόφερ, έχει το λόγο. Και σου δίνω 15 λεπτά ε, να τηρηθούν. Ευχαριστώ. To talk about για να μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό θέμα, η βία κατά των γυναικών και η φτώχεια. Το όνομά μου είναι Ραγκίνα Πόφερ και εργάζομαι για τον οργανισμό Γυναίκε Κατά τη Βία στην BRIF στην Ευρώπη. Είναι δίκτυο ε, γυναικών που καταπολεμούν την ανισορροπία εναντίον του. Ιδρύθηκε το 1994 και λειτουργεί μεταξύ από 91 εστιακών σημείων σε 47 ευρωπαϊκές χώρες. Το δίκτυο WAVE ε, έχει περίπου 4.000 κυβερνητικέ οργανώσει όπω το Women's Shelter, Women's Helpline και διάφορα κέντρα παροχή συμβουλών. Και συντονίζεται το δίκτυο μέσω τη υπηρεσία του γραφείου ε, WAVE που είναι εδρεύει στη Βιέννη. Και το γραφείο αυτό έχει διενεργήσει αρκετά προγράμματα, εφαρμόσει αρκετά προγράμματα Δάφνη και παίρνει χρηματοδότηση από τις χορηγίες Δάφνη. Το σημερινό θέμα είναι πώς η φτώχεια επηρεάζει τις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την κοινή έκθεση για την κοινωνική ένταξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, βλέπουμε ότι υπάρχει πολυσχηδής ορισμός της φτώχειας. Θέλουμε να μειώσουμε και περιορίζουμε συνήθως εκεί τη φτώχεια στα χαμηλά εισοδήματα και στους χαμηλούς πόρους. Η φτώχεια όμως είναι πολλαπλό μειονέκτημα. Ανεργία, χαμηλό εισόδημα, κακή στέγαση, ανεπαρκής πρόνοια, ε, εκτός διαβίου εκμάθησης, αποκλεισμός, περιθωριακή, μπαίνει στο περιθώριο σαν φάσει συμμετοχή στην πολιτική, στον πολιτισμό κλπ. Και δύσκολο να απολαμβάνει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θέλω να αξιολογήσω την ε, κατάσταση των γυναικών όσον αφορά τη βία που ασκείται εναντίον τους. Η φτώχεια και η εξάρτηση είναι ε, παράγοντε κινδύνου που οδηγούν στη βία. Γυναίκες και παιδιά που έχουν μια, ζουν σε βίαιη σχέση μπαίνουν σε πολλές παγίδες από φτώχεια. Και δεν μπορούν να αφήσουν αυτή τη βία σχέση και να ζήσουν ε, τη ζωή ε, κανονικά, χωρίς βία, να ξεφύγουν. Είναι δύσκολο να ξεφύγουν άμα είναι φτωχοί. Και οι γυναίκες παιδιά τους είναι πιο ευάλωτοι στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Κυρίω οι μετανάστριες γυναίκες ε, με αναπηρία και ηλικιωμένες γυναίκες που είναι θύματα βίας. Πέρα των παγίδων φτώχειας που αντιμετωπίζονται, μέσω αυτής της βίας σχέσης αντιμετωπίζουν αυτές τις παγίδες οι γυναίκες, υποφέρουν και από διάκριση, πολλαπλή διάκριση και εξαρτώνται όλο και περισσότερο λόγω ε, δομικής ανισότητας, ανίσων ευκαιριών γλωσσικών φραγμών και προβλημάτων επικοινωνία. Έχουν και αυτά τα προβλήματα από πάνω. Και άλλος ένας λόγος που είναι σημαντικό στη η κατάσταση είναι και ο Το θέμα αυτό εξαιρείται από τη συζήτηση περί φτώχειας. Η φτώχεια των γυναικών εξετάζεται οριζόντια, στο περιθώριο και σχέση μεταξύ βίας και γυναικών και φτώχειας δεν εξετάζεται. Σχεδόν καθόλου. Υπάρχει και μεγάλη έλλειψη στοιχείων. Το ξέρουμε αυτό όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών. Και δεν εκπροσωπούνται επακριβώς τα στοιχεία για τη φτώχεια γυναίκες. Η χρήση των οικιακών εισοδημάτων σαν βάση μέτρησης των στατιστικών στοιχείων για τη φτώχεια, υποθέτουμε ότι κάθε τέλο στην οικογένεια παίρνει τα ίδια χρήματα. Οι γυναίκες πολύ συχνά δεν ελέγχουν τα εισοδήματά τους. Πιο συχνά το χαμηλό εισόδημα των γυναικών ξοδεύεται για τα παιδιά και άλλα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας. Η σχέση μεταξύ βίας γυναικών και φτώχειας δεν εξετάζεται, δεν λέμε αντιπόψη στα στατιστικά στοιχεία επαρκώς. Το ίδιο ισχύει πάρα πολύ συχνά στι στρατηγικές, πολιτικέ και διάφορα σχετικά έγγραφα. Τα περισσότερα εθνικά σχέδια δράση όσον αφορά την κοινωνική ένταξη δεν έχουν οπτική γωνία των δύο φύλων και αγνοούν τι γυναίκε συχνά. Η βία και η φτώχεια που σχετίζονται είναι κάτι που δεν λαμβάνεται υπόψη ο σχετισμό του. Και ευάλωτε ομάδε γυναικών όπω είναι οι μετανάστε, οι γυναίκε με αναπηρίε και οι ηλικιωμένε που είναι θύματα βία εξετάζονται ακόμα λιγότερο αυτές τις κατηγορίες που πανέφερα οι τρεις. Έτσι περαιτέρω, η οργάνωσή μας που υποστηρίζει τις γυναίκες που επιβιώνουν από τη βία, βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να συμβάλλουμε στη σύνταξη τέτοιων εγγράφων διάμορφης πολιτικής σαν οργανισμοί. Είτε διότι μας λείπουν πόροι, είτε γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη η δική τους οπτική γωνία θεωρούμε ότι η βία κατά των γυναικών και η φτώχεια εκφράζουν δομική βία και τα δύο αυτά στοιχεία. Ο τίτλος του πάνελ είναι «Οι διαστάσεις της φτώχειας που πλήττει τις γυναίκες, οι γυναίκες που επιβιώνουν από τη βία και η βία κατά των παιδιών». Σχετικά με όλα αυτά, η βία κατά των γυναικών είναι η πιο συχνή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη σημερινή εποχή. Αν δείτε τα στοιχεία, βλέπετε το 1 πέμπτο μέχρι 1 τέταρτο των γυναικών που ζουν στην Ευρώπη υπήρξαν θύματα φυσικής βίας τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Τι σημαίνει αυτό. 100 εκατομμύρια γυναίκες από 500 εκατομμύρια πληθυσμό που ζουν σε 27 ευρωπαϊκά κράτη-μέλη πλήττονται από τη βία. Και όσον αφορά τη βία που ασκείται από το σύντροφο, συμπεριλαμβάνονται πάντα και τα παιδιά. Είτε παθητικά είτε ενεργά. Είναι θύματα παθητικής ή ενεργού βίας τα παιδιά. Το 2008 και 2009 μαζί με τους την Oxfam του Ηνωμένου Βασιλείου και Λαμόρε της Ιταλίας ετοιμάσαμε ανακοίνωση για την σώτα των φίλων και πώς λαμβάνεται υπόψη αυτή η διάσταση διαμόρφωση των πολιτικών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από το πρόγραμμα δράσης Progress και ήταν τα καθήκοντα του WAVE να εντοπίσουμε τους κινδύνους που δημιουργούνται από τη φτώχεια και που δημιουργούν βία κατά των γυναικών. Είδαμε ότι η βία και η φτώχεια βασίζονται στην δομική βία. Και υπάρχουν παγίδες φτώχειας για τις γυναίκες θύματα της βίας. Πρέπει να εντοπιστούν στο κοινωνικοπολιτικό ε, επίπεδο και στις κοινωνικές δομές. Στην ε, παιδεία, στην πρόνοια, στην οικονομία, στα, στα κοινωνικά επιδόματα και στο νομικό σύστημα πρέπει όλα αυτά να λαμβάνονται υπόψη. Στο πρόγραμμα αναλύσαμε την κατάσταση. Είδαμε τι γίνεται στην Αυστρία. Τα αποτελέσματα σε αυτή την έκθεση που βλέπετε. Εδώ εντοπίζεται η φτώχεια, οι παγίδες φτώχειας και έχουμε και συστάσεις τι μπορεί να βελτιωθεί. Για να βελτιωθεί η κατάσταση για τις γυναίκες που έχουν επιβιώσει κρούσματα βίας, από κρούσματα βίας μάλλον. Λοιπόν, γενικά, ποιο ήταν το σημαντικό που είδαμε. Ότι οι γυναίκες που έχουν επιβιώσει από κρούσματα βίας δεν επηρεάζονται μόνο από μία από ένα κρούσμα φτώχεια, ένα σύμπτωμα φτώχεια, μια παγίδα φτώχεια. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι από τη φτώχεια. Πολλέ παγίδε δημιουργούνται από τη φτώχεια. Φυσική, σεξουαλική, ψυχολογική βία δημιουργεί προβλήματα υγεία. Τα προβλήματα υγεία δεν κοστίζουν μόνο πόνο στι γυναίκε, αλλά αυξάνουν και τον κίνδυνο να χάσει η γυναίκα τη δουλειά τη. Γιατί λόγω απουσίας, λόγω άδειας ασθενείας και μειωμένης απόδοση στη δουλειά. Πέραν αυτού, τα προβλήματα υγείας αυξάνουν το κόστος της και περίθαλψης και λοιπά. Οι μετανάστριες, παραδείγματος χάρη, πολύ συχνά δεν εργάζονται και δεν έχουν δική τους ασφάλιση. Εάν μια μετανάστε αποφασίσει να φύγει από τον βίο σύντροφό της, δεν έχει κάλυψη υγείας. Πιο πέρα. Οι γυναίκες θύματα βίας πολύ συχνά εξαιρούνται από προγράμματα περαιτέρω κατάρτισης και εκπαίδευσης. Είτε λόγω οικονομικής βίας, βλέπετε δεν έχουν τα χρήματα για να πληρώσουν για την κατάρτιση, οι μετανάστες έχουν και το εξή πρόβλημα. Δεν έχουν προσόντα. Προσόντα που απέκτησαν στη χώρα προέλευσής τους δεν αναγνωρίζονται στη χώρα υποδοχής. Και γι' αυτό πολύ συχνά δέχονται δουλειές που δεν ανταποκρίνονται στα προσόντα τους. Ξέρουμε όλοι τα προβλήματα αυτά. Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν τη δουλειά, πολλές γυναίκες θύματα βίας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Διότι έχουν πρόβλημα με την περίθαψη τη μέρη των παιδιών. Αυτοί που βιοπραγούν εναντίον τους πολύ συχνά δεν τους επιτρέπουν τη να το, να μάλλον να ασκήσουν κάποιο επάγγελμα. Οι μετανάστρες κυρίως είναι ιδιαίτερα ευάλωτε. Γιατί? Διότι συχνά δεν έχουν άδεια εργασία. Αυξάνει περισσότερο κίνδυνος φτώχειας όταν οι γυναίκες έχουν το θάρρος να εγκαταλείψουν το βίο σύντροφό τους διότι πολύ συχνά πρέπει να φύγουν από το σπίτι τους, από το διαμέρισμά τους, να γίνουν άστεγες, χάνουν και τη δουλειά τους, γιατί είναι επικίνδυνο να πάνε στη δουλειά τους, χάνουν επίσης την άδεια διαμονής τους και πολλές γυναίκες γίνονται μητέρες, ε, δημιουργούν μια μονογονική οικογένεια γιατί δεν είναι ο άλλος γονέας πλέον μαζί τους. Η μόνη λύση που έχουν αυτές οι γυναίκες είναι να πάνε σε ένα καταφύγιο γυναικών. Και βλέπουμε ότι το καταφύγιο γυναικών είναι κάτι καλό. Αποφεύγουμε έτσι την άσκηση βίας κατά των γυναικών και προστατεύουμε τις γυναίκες και όχι μόνο από τη βία αλλά και από τη φτώχεια. Τα καταφύγια των γυναικών προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Για όλες τις ε, γυναίκες, δωρεάν. εξετάζουν τι γίνεται και με τι ευάλωτε γυναίκε, μετανάστριε, γυναίκε με αναπηρίε, ηλικιωμένε γυναίκε. Λαμβάνουν υπόψη τι ειδικέ ανάγκε των ευάλωτων ομάδων. Αυτή η ειδική υπηρεσία προσπαθεί να απελευθερώσει τι γυναίκε από εξάρτηση. Ακολουθείται μια σφαιρική προσέγγιση, ολιστική. Σε ένα καταφύγιο γυναικών, οι γυναίκε υποστηρίζονται. Του βοηθά να βρουν τη σωστή δουλειά. Του βοηθούν να βρουν ε, κατοικία ένα διαμέρισμα. Παίρνουν ειδικέ συμβουλέ. Οι γυναίκε που έχουν, τα παιδιά μάλλον που έχουν πληγεί από βία, παίρνουν ειδικέ συμβουλέ. Και τα καταφύγια γυναικών παρέχουν και νομική αρρωγή, ψυχολογική στήριξη κατά τη διάρκεια δικασίας, ε, και κατά τη διάρκεια εκδίκαση τη υπόθεσή του. Υποστηρίζουν τι γυναίκε στην ιατρική περίθαλψη που χρειάζονται κλπ. Τα τελευταία χρόνια πετύχαμε μεγάλη πρόοδο όσον αφορά την νομοθεσία. Είναι σημαντικότατο κάθε θύμα βίας να έχει δικαίωμα προστασίας, δικαίωμα υποστήριξης. Όταν είναι θύματα βίας, όπως σας είπα. Όμως, πέρα από την νομοθεσία, είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρέχονται αρκετές υπηρεσίες, να υποστηρίζονται οι γυναίκες θύματα βίας. Πολλές οργανώσεις γυναικών δεν έχουν χρήματα, αρκετά χρήματα. Γι' αυτό δεν μπορούν να πετύχουν τις υπηρεσίες τις ενδεδειγμένες για τα θύματα βίας της γυναίκε σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Γι' αυτό συστήνουμε ένθερμα να υποστηριχθεί η τεχνογνωσία των μη κυβερνητικών οργανώσεων γυναικών όσον αφορά τη φτώχεια και τη βία όμως. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να υπογραμμίσω ότι είμαστε ανοιχτές και στο ότι χρειάζεται μια σωστή συνεργασία και με οργανισμούς έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξανά σας ευχαριστώ κυρία Βουέμπχόφερ λοιπόν. Τώρα θα καλωσορίσω εδώ στη συζήτηση την κυρία Μαρία Λία Ποπ που είναι καθηγήτρια ε, πρίτανης στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών και σε σπουδές που έχουν να κάνουν με τα μέσα μαζικών ενημέρωσης στην Οραντέα από στη Ρουμανία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, είναι μεγάλη μου τιμή που παρευρίσκομαι εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το θάρρος που επιδείξατε να καλέσετε κάποιον από την Ανατολική Ευρώπη. Η δική μου παρουσίαση θα γίνει στα ρουμανικά. Θα προσπαθήσω λοιπόν να βάλω σε λειτουργία εδώ ε, το μηχάνημα. Δεν είμαι πολύ καλή σε αυτά, αλλά θα προσπαθήσω. It's low battery.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 doesn't allow me to to have a Okay. I will ask for the permission to uh, speak in my mother tongue because my English is very limited, so I, I can. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να μιλήσω στην μητρική μου γλώσσα γιατί τα αγγλικά μου είναι περιορισμένα.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 εδώ στο χάρτη βλέπουμε την κατάσταση των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς υπάρχει και πάλι ένα τεχνικό πρόβλημα με τη διερμηνία. Δεν υπάρχει μετάφραση από τα ρουμανικά. Okay. In English, In English. Problem with translation. Okay. Anyway, Μπορείτε να δείτε το χάρτη. Και μπορείτε να δείτε τις ε, περιοχές όπου είναι ιδιαίτερως έντονο το φαινόμενο της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο χάρτη το βλέπουμε με χρώμα γκρι. Ζητώ συγγνώμη για τα αγγλικά μου, λέει η μιλήτρια τα επίπεδα φτώχειας το 2007. Το βλέπουμε εδώ στη διαφάνεια. Εάν δούμε λοιπόν τα στατιστικά στοιχεία, εάν τα εξετάσουμε προσεκτικά, μπορούμε να προβλέψουμε την ε, κρίση. Εάν η φτώχεια επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες στην Ανατολική Ευρώπη, το κατά πόσο τις επηρεάζει περισσότερο στην Ανατολική Ευρώπη ή όχι, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα με απασχολήσει στην παρουσίασή μου. Η απάντηση είναι και ναι και όχι. Δηλαδή, ναι, επηρεάζει καταρχήν περισσότερο τις γυναίκες στο ανατολικό τμήμα τη Ευρώπης, ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι σε επηρεάζει Μπορώ να συνεχίσω τη μητρική μου γλώσσα, λέει η ομιλήτρια. Όχι στα αγγλικά, παρακαλώ, λέει η πρόεδρος. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να με καταλάβετε στα αγγλικά. Γίνει πάλι μια προσπάθεια στα ρουμανικά, να δούμε αν λειτουργεί η διερμηνία. Ευχαριστώ mai sunt zone sorry for, uh, sunt acolo că Υπάρχουν άλλες ε, περιοχές ε, φτώχειας. Υπάρχουν άλλες ζώνες φτώχειας και οι ζώνες αυτές που έχουν καταδικαστεί στη φτώχεια είναι οι περιοχές της υπαίθρου στην Ανατολική Ευρώπη. Οι ζώνες συγκέντρωσης της ε, φτώχειας, της μεγάλη πόλη υφίστανται επίση ιδιαίτερα ε, στις παρυφές των πόλεων, εκεί όπου ζουν περισσότεροι φτωχοί.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 I'm so sorry. I'm real sorry, but now there are translation problem again. So if possible, if you could continue in English. Σας παρακαλούμε, λέει η Πρόεδρος, μήπως μπορείτε στα αγγλικά παρόλα αυτά. Τέλος. Please. There is no translation problem. In English.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 Listen now, information about translation. Θα ήθελα να σας μια πληροφορία σχετικά με την ε, διερμηνία. From From Δεν υπάρχει, λέει, η δυνατότητα προς τα γαλλικά από τα ρωμανικά, αλλά σε όλες τις άλλες μπορούμε να έχουμε από τα ρωμανικά, ε, ρουμανικά συγγνώμη, προς τα γαλλικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό τώρα. Εγώ λοιπόν στα γερμανικά στα τρία, στο το κανάλι 3 μπορούμε να έχουμε προς τα γερμανικά. Άρα μπορούμε να συνεχίσουμε ε, και ελπίζω να συνεχίσουμε τώρα χωρίς να έχουμε ξανά κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Παρακαλώ λέει ο Πρόεδρος. Κύριε πο Γεια, ξαναπροσπαθήστε. Συγγνώμη, λέμε μιλήτε, δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω στα γαλλικά. Λοιπόν, πρόκειται για αυτές τις ζώνες όπου ζουν περισσότερες μετανάστριες. Αυτές είναι οι ζώνες φτώχειας της μεγάλης πόλης. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι η φτώχεια στην υπεθρεφική διαστάση που δεν μπορούμε καν να τις συνδιανοηθούμε. Για να απαντήσουμε λοιπόν την, το ερώτημα σε σχέση με το τρόπο που επιβαρύνει η φτώχεια της γυναίκες, θα πρέπει να πούμε ότι δεν πλήττονται, δεν υποφέρουν όλες οι γυναίκες στην Ανατολική Ευρώπη. Εάν δούμε και πάλι το χάρτη, θα καταλάβουμε ότι η φτώχεια δεν είναι τόσο μεγάλη στην Πολωνία, είναι περιορισμένη στη Δημοκρατία της Τσεχίας, είναι σχετικά περιορισμένη στην Αυστρία, την Ουγγαρία κλπ. Δεν υπάρχει λοιπόν τόσο εκτεταμένη φτώχεια στις ε, περιοχές αυτές, όσο στις περιοχές που, είναι, που έχουν τη σήμανση με τον γκρι χρώμα στη διαφάνεια. Μπορούμε, ε, κατανοούμε λοιπόν ότι η φτώχεια έχει μια γεωγραφική διάσταση. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι η φτώχεια κατ' ουσία συνδέεται με το φύλλο. Στην ε, πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών μελών 17% των γυναικών είναι σε κατάσταση φτώχειας, δηλαδή πάνω από μία στις πέντε γυναίκες. Με άλλα λόγια, υπάρχουν περισσότερες γυναίκες που ζουν ε, μέσα στη φτώχεια από ότι άνδρες. Στους άνδρες το αντίστοιχο ποσοστό είναι ένα στους 7. Όταν ε, δούμε τα μονογονεϊκά σχήματα, εδώ 35% ε, των γυναικών αυτών σε μονογονεϊκές οικογένειες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Για... Ε, και πολύ συχνά τα επιδόματα για τα παιδιά είναι περιορισμένα και πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της ε, μητρικής ε, άδειας, της άδειας του τοκετού μάλλον, οι γυναίκες είχαν εντελώς τα, τις αποδοχές τους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια περιοχή του κόσμου με έναν ε, πληθυσμό που γυράσκει όλο και περισσότερο. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν νέους ε, Ευρωπαίους πολίτες που να εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη εξέλιξη. Και από την άλλη ε, χρησιμοποιούμε όμως ένα κοινωνικό μοντέλο το οποίο τιμωρεί τη μητρότητα. Στο παρελθόν οι γυναίκες υπέφεραν, οι μητέρες υπέφεραν λιγότερο. Γίνεται συχνά, λέγεται συχνά ότι οι μητέρες ότι οι γυναίκες δεν υποφέρουν όσο οι άνδρες από την κρίση. Γιατί οι πρώτες ζώνες ε, που πλήττονται από μια κρίση, από μια βιομηχανική κρίση, είναι οι άνδρες. Τα πρώτα είναι οι άνδρες. Γιατί αυτοί πλήττονται περισσότερο στις θέσεις εργασίας τους. Ωστόσο τώρα η κρίση γενικεύεται και θα έχει δυσμενέστερες επιπτώσεις για τις γυναίκες. Για τις ε, γυναίκες υπαλλήλου ε, διαπιστώνεται μία συρρήκνωση των θέσεων εργασίας. Επίσης υπάρχουν όλο και λιγότερες θέσεις εργασίας τα κομμωτήρια για παράδειγμα ή στα Ινστιτούτα Αισθητικής. Δηλαδή, πάρα πολλέ γυναίκε τα επόμενα χρόνια θα χάσουν τι θέσει εργασία τους. 12 χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε 12 χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν ε, οι γυναίκε σε μια κατάσταση ανεργία που τι πλήττει πολύ περισσότερο από τον ανδρικό πληθυσμό. Ο κίνδυνος να απολέσουν τη θέση εργασία του είναι μεγαλύτερο για τι γυναίκε από ό,τι για του άνδρες στο σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. 17% των γυναικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβίουν σε συνθήκες φτώχειας, 17% επαναλαμβάνω, και έχουν ελάχιστες ε, αποδοχές που είναι κάτω από το 70% του, του εθνικού κατακεφαλήν εισοδήματος. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι στο Λουξεμβούργο οι γυναίκες έχουν ελάχιστες αποδοχές που είναι κάτω από τα 1641 ευρώ. Στη Βουλγαρία αυτές οι ελάχιστες ποδοστές είναι 123 ευρώ το μήνα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμούμε να μειώσουμε την φτώχεια των γυναικών μέσω μιας ανακατανομής. οι χώρες που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια, κάτω από τις συνθήκες της παρούσας κρίσης, είναι οι γυναίκες στη Ρουμανία, στις χώρες της Βαλτικής, στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την ε, Πορτογαλία. Ε, δηλαδή στις, ε, περιφερειακές, στις χώρες της περιφέρειας. Αυτές είναι οι διαστάσεις της φτώχειας στη βάση των ε, στατιστικών ε, στοιχείων. Η φτώχεια όμως ε, παρουσιάζει και ένα κοινωνικό πρόβλημα. και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να την ε, περιγράψουμε τη φτώχεια με κοινωνικοψυχολογικούς όρους ή από τη σκοπιά της κοινωνικής πολιτικής. Και υπό την έννοια αυτή θα ήθελα να σας προτείνω ορισμένους ε, ε, ορισμούς της φτώχειας. Θα ήθελα να με συγχωρήσετε, λέει η ομιλήτρια, δεν είχα φορέσει τα γυαλιά μου προηγουμένως και παρέλειψα να σας αναφέρω κάτι το οποίο όμως είναι στοιχείο, είναι σημαντικό στοιχείο. Η φτώχεια μπορεί να περιγραφεί επίσης με όρους γενεάς, γιατί δεν είναι εξίσου φτωχές όλες οι γενιές. Όπως είπε και συνάδελφός μου η κυρία Βεπχόφερ, οι νεαρές γυναίκες Καθώ και οι γυναίκε μεγαλύτερη ηλικία είναι ιδιαίτερα φτωχέ, ή πιο φτωχέ σε σχέση με τον ενεργό γυναικείο πληθυσμό. Και υπάρχει και μια άλλη διάσταση της ε, φτώχειας, η οποία επίση θα μπορούσε να εμφανιστεί με στατιστικά στοιχεία, δηλαδή στη ε, βάση του έτους γέννησης. Οι νεαρές γυναίκες οι ευθείε πρέπει καταρχήν να εισέλθουν στην αγορά εργασία είναι ιδιαίτερε στοχές, το ίδιο όπως και οι γυναίκες που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Οι νεαρές γυναίκες δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν πλέον μια θέση εργασία και αυτή η θέση εργασία πολύ συχνά βρίσκεται σε μια γκρίζα ζώνη. Ε, ορισμένοι κοινωνιολόγοι συνάδελφοί μου μου είπαν ότι στην Νότια Ιταλία είναι ιδιαίτερος δύσκολο για μια γυναίκα με ακαδημαϊκή μόρφωση, με πτυχίο, να βρει μια θέση εργασίας. Είναι πολύ πιο δύσκολο μια γυναίκα που έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο να βρει μια θέση εργασίας από μια γυναίκα που δεν έχει τόσο υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Εκείνες οι γυναίκες που βρίσκουν τελικά μια θέση εργασίας βρίσκουν κακά αμοιβόμενε θέσει εργασία που βρίσκονται αυτήν ακριβώ σε αυτή την κρίζα ζώνη τη αγορά. Μία γραμματέα ε, μπορεί να κερδίσει χίλια ευρώ ή μάλλον τις υπόσχονται ε, χίλια ευρώ το μήνα ως μισθό, αλλά στην ουσία παίρνει 500 ευρώ και δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Ή μια νερή γυναίκα Ρώμα, τσιγκάνα, ή οι γυναίκες ή οι γυναίκες που είναι άρρωστες ή έχουν μικρά παιδιά, αυτές είναι οι πιο φτωχές κατηγορίες γυναικών στην Ευρώπη. Ε, μητέρες ε, παιδιών με χρόνιες παθήσεις ή μητέρες παιδιών με αναπηρίες ε, βρίσκονται πραγματικά σε μια απελπιστική κατάσταση και δεν έχουν καμία ειδική υποστήριξη. Γυναίκες σε μονογονεϊκές οικογένειες που ακόμα σπουδάζουν εντάσσεται στις κατηγορίες των φτωχών γυναικών. Στην Πολωνία υπάρχουν ιδιαίτερες κατηγορίες με teenager νερών γυναικών που είναι έγκυες. Και επίσης γυναίκες πάνω από τα 55 βρίσκονται επίσης σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου. Ε, προσπάθησα ε, ή μάλλον θα ήθελα να σα καταγραφήσω τρία πορτρέτα γυναικών που ζουν σε συνθήκε φτώχεια. Μία γυναίκα από την Πολωνία, η Άννα, 19 ετών, φοιτήτρια και έγκυο. Η οποία δυστυχώ είναι αναγκασμένη να εγκαταλείψει τι σπουδέ τη και να παντρευτεί για να μπορέσει να μεγαλώσει το παιδί στου κόλπου μια οικογένεια. Μία άλλη ε, γυναίκα από τη Ρουμανία, 28 ετών, η οποία δεν μπορεί να παντρευτεί. Ή μία γυναίκα από 60 ετών από την Ισπανία, η οποία δεν μπορεί πλέον να πληρώσει το νίκη για το σπίτι της και ε, πήγε σε ένα ίδρυμα για να διαμείνει εκεί, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα έξοδα. Βεβαίω για να κατανοήσουμε την κατάσταση αυτών των γεγονότων χρειαζόμαστε περισσότερα κοινωνικά και ψυχολογικά στοιχεία. Θα ήθελα να πω ε, περισσότερα πράγματα σαν ένα ψυχολογικό πορτρέτο της φτώχειας. Υπάρχει η λεγόμενη πυραμίδα Μάσλο, η οποία ε, αφορά πέντε επίπεδα αναγκών. Το βασικό επίπεδο αφορά ε, την στέγαση, την τροφή και την ένδυση. Όταν μιλάμε για τη φτώχεια, μιλούμε συνήθως, αναφερόμαστε συνήθως μόνο σε αυτά τα τρία στοιχεία, αλλά υπάρχουν και άλλα επίπεδα που τελικά οδηγούν τις γυναίκες στην απελπισία. Άλλα στοιχεία που οδηγούν τις γυναίκες στην απελπισία. Ε, θα πρέπει να κλείσω κάπου την ομιλία μου εδώ είδαμε ένα χάρτη κατανομής της ε, φτώχειας διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μπορούμε να τη συγκρίνουμε με τη διαφάνεια που σας έδειξα στην αρχή, γιατί υπάρχει μια σχέση μεταξύ της φτώχειας των γυναικών και της εκπροσώπησης των γυναικών. Ποια είναι η προτεραιότητα που θα πρέπει να έχει ο αγώνας κατά της ε, φτώχειας. Θα πρέπει να υπάρξει μια υποστήριξη των γυναικών και μια επίδειξη αλληλεγγύης προς τις γυναίκες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τώρα, κάποια συμπεράσματα λέει η ομιλήτρια. Η φτώχεια θα πρέπει να προσλεφθεί στις τρεις της διαστάσεις, τη γεωγραφική, τη διάσταση του φύλου και των γενεών και Επίσης ε, τη διάσταση ε, της ηλικίας. Πολύ συχνά η φτώχεια μας μπορεί να προσλάβει ένα πραγματικά ε, καταστροφικό χαρακτήρα. Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι η φτώχεια είναι ιδιαίτερα σοβαρό φαινόμενο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αφήσουμε τη μοίρα των γυναικών στα χέρια των αντρών και θα ήθελα να διβάσω το μήνυμα αυτό σε όλες τις γυναίκες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λέγοντας ότι οι γυναίκες στη Ρουμανία εμπιστεύονται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ελπίζουν ολοντικά μια...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 Τώρα θα δώσουμε, λέει, το λόγο στους συναδέλφους και εξή να είσαστε σύντομοι, σύντομες, δύο-τρία λεπτά, γιατί είχαμε και όλες αυτές τις καθυρίσεις λόγω των τεχνικών προβλημάτων. Πρώτα, λοιπόν, θα δώσω το λόγο στην κυρία Καμπριέλ Τσίμερ, η οποία είναι συγγήτρια από την Επιτροπή Απασχόλησης και μέλος της ΓΚΟΕ, της Ευρωπαϊκής Αριστερής Ομάδας, Παρακαλώ, κυρία Ζήμερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να συμμετάσχω σε αυτή την ε, ακρόαση ως εκπρόσωπης της Επιτροπής Απασχόλησης και ταυτόχρονα θα ήθελα να παρουσιάσω ορισμένες ε, πτυχές ε, ε, τις οποίες, ε, του φαινομένου τις οποίες επεξεργάζομαι εγώ στο πλαίσιο της εργασίας μου και της εκπόνησης της δικής μου έκθεσης. Θα ήθελα να αναφέρω εισαγωγικά δύο παρατηρήσεις γενική φύσεως που είναι σημαντικές όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της φτώχειας στις γυναίκες. Καταρχήν, ε, αφορά το ατομικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να μπορεί να διαβεί σε αξιοπρεπείς συνθήκες και να έχει πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Αυτό αφορά τόσο τις γυναίκες όσο και τα ανθρώπινα όντα, αλλά και ειδικότερα τις γυναίκες ως συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα του πληθυσμού. Η δεύτερη παρατήρηση έχει ω εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του αγώνα για την ε, ίση αντιμετώπιση των δύο φύλων τάσεται υπέρ της απαγόρευσης ε, των ε, διακρίσεων. Ωστόσο όλοι γνωρίζουμε ότι και στις δικές μας χώρες υπάρχουν ορισμένοι που εκμεταλλεύονται την προσπάθεια αυτή που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε κάποιες άλλες χώρες όπως είναι η Σουηδία. Ο αγώνας για την συμμεταχείριση των δύο φύλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο των χωρών μελών προσκρούει σε υπερβολικά στενά όρια όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη δεν επιδεικνύουν το ίδιο επίπεδο δέσμευσης ε, για τον αγώνα, στο πλαίσιο του αγώνα για την καταπολέμηση της φτώχειας. οι διακρίσεις κατά των γυναικών δεν καταργούνται όταν οι άνδρες και οι γυναίκες είναι εξίσου φτωχοί και ζουν σε κοινωνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Και θα ήθελα να σας εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. Ως βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσπαθήσουμε ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπονήσει κοινέ στρατηγικές και κοινούς, να δεσμευτεί στους κοινούς στόχους στο πλαίσιο του αγώνα για την καταπολέμηση της φτώχειας, ιδιαίτερα όσον αφορά ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, γυναίκες, παιδιά, ε, μέλη εθνοτικών ε, μειονοτήτων, μετανάστες κλπ. Ο στόχος της στρατηγικής 2020, ε, η στόχη δεν είναι επαρκής. Το να βγάλει κανείς 20 εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια, αυτός είναι ελλειπής στόχος εάν δούμε ότι υπάρχουν 80 ή 90 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν επισήμω κάτω από το όριο τη φτώχεια. Ε, και είναι και λυπή τα στοιχεία για του αφορά του Ρωμά, τι αφρονικέ μειονότητε, του μετανάστε κλπ. Άνθρωποι που δεν ε, μπαίνουν καν, δεν καλύπτονται καν από τι στατιστικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ίδιο ισχύει και για τα 19 εκατομμύρια παιδιά. Με αυτό θα ήθελα να σα επισημάνω ότι προσπαθώ να τονίσω αυτό στη δική μου έκθεση, γιατί θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα προβληματικό το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το θέρος αυτού του έτου, δημιούργησε τελικά ε, μία, ένα πρόσχημα για τη συγκάλυψη της φτώχειας. Εάν ε, θέλουμε να υπάρξει μία κοινή στρατηγική, θα πρέπει να μπορούμε να συγκρίνουμε σωστά την κατάσταση που επικρατεί στι διαφορέ χώρε Και πραγματικά έχετε δίκιο ε, να πείτε ε, ότι στην Ανατολική Ευρώπη η φτώχεια προσλαμβάνει εντελώ διαφορετικέ διαστάσει από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη και θα πρέπει να κάνουμε εδώ μια διαφοροποίηση. Από το 1995, και θα ήθελα να σα επιστήσω γιατί το θεωρώ σημαντικό. Από το 1995 η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έθεσε το σχετικό όριο απειλής από τη φτώχεια. Δηλαδή 16% του, ε, του εθνικού προϊόντος, του εθνικού κατακεφαλήν εισοδήματος. Και εδώ έχουν προσθεθεί δύο άλλοι δείκτες που θεωρώ ότι είναι σωστοί. Ε, κάποιες δυσκολίες όσον αφορά την εξασφάλιση αγαθών ή υπηρεσιών και ο δεύτερος δείκτης είναι η μακροπρόθεσμη ανεργία εντό τη οικογένεια. Το πρόβλημα όμω έγκυται στο εξή και θα ήθελα να σα επιστήσω την προσοχή. Οι χώρε έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τους δικούς τους δείκτες και με τον τρόπο αυτό τελικά ε, παρακάμπτεται η δυνατότητα εκπόνησης μιας κοινή στρατηγικής. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στη Φρασίσκα Μπράτνε που είναι σκιώδης εισηγήτρια στην ομάδα των Πρασίρων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. <coughs> Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τις κυρίες που έκανε τις παρουσιάσεις. σχολιά σου, εν συντομία κάποια σχόλια. Συμφωνώ με τα περισσότερα που υπόθηκαν από τις δύο προλαλήσεις Νομίζω ότι θα πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα από την πτυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό έχει ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαίωμα κάθε γυναίκας που πρέπει να έχει τα ίδια κοινωνικά δικαιώματα. Και τα κορίτσια επίσης και υπάρχει έλλειψη ορατότητας, θεωρώ, στην Ευρώπη όσον αφορά τη φτώχεια των γυναικών και τον κοινωνικό του αποκλεισμό και θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη μονάδα κάθε νοικοκυριού που καθορίζει το εισόδημα για καθοριστή φτώχεια και θεωρεί ότι σώτιμα κατανέμονται τα εισόδηματα στα νοικοκυριά. Το βρίσκω ενδιαφέρον. Πολύ συχνά βλέπουμε κατά νοικοκυριό τι γίνεται και υποθέτουμε ότι το εισόδημα μοιράζεται ισότιμα μεταξύ ανδρών και γυναικών και συνήθως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και επισκιάζει την φτώχεια των γυναικών κατά πολύ και εντό των οικοκυριών αυτή η προσέγγιση. Θα πρέπει εκεί να επεξεργαστούμε την ορατότητα, να αναθεωρήσουμε το πώ προσμετρούμε το εισόδημα του νοικοκυριού. Και βεβαίω και η ορατότητα τη θηλυκή φτώχεια ξεπερνά αυτό το όριο. Πολύ δουλειά χρειάζεται να γίνει. Στη Γερμανία, παραδείγματι, η ομάδα των μητέρων που εκπαιδεύουν μόνες τους τα παιδιά αντιμετωπίζουν μεγάλο κίνδυνο φτώχειας και είναι λυπηρό αυτό. Εκείνες που έχουν μεγάλο βάρος και το φέρουν για όλη την ε, κοινωνία αυτό το βάρος να αντιμετωπίσουν το μεγαλύτερο κίνδυνο για τη φτώχεια. Οπότε έρχομαι σε κάτι που έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση. Οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα σε δικαιώματα όσον αφορά κοινωνική προστασία, φορολόγηση, επιδόματα. Το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας θα πρέπει να τους καλύπτει, κυρίως τα συντοξιδοτικά, να καλύπτονται εκεί τα δικαιώματα των γυναικών. Να μην αντιμετωπίσουν τη φτώχεια από τη στιγμή που σταματούν να δουλεύουν ή όταν χειρεύσουν ή όταν ε, μείνουν μόνες ή πάρουν διαζύγιο. Και τα ατομικά δικαιώματα, η ίδια ιδέα αφορά και το άσυλο. Και άλλα προβλήματα. Εκείνες που μπήκαν σε μια χώρα έχοντας παντρευτεί κάποιον Χρειάζεται να τονίσουμε, γραμμίσουμε τα ατομικά δικαιώματα των γυναικών. Και κάτι άλλο που είναι κρίσιμο. Ποιότητα μέρημνας, προσβάσιμη μέρημνα, φθηνή μέρημνα. όχι μόνο για τα παιδιά, για τη μέρημνα για τα παιδιά, αλλά και μέρημνα εξαρτωμένων ανθρώπων, ηλικιωμένου και άλλα μέλη του νοικοκυριού. Τέλος. Η διαφορά αμοιβή μεταξύ των δύο φύλων. Έχει συζητηθεί αρκετά το θέμα αυτό. Και κλείνοντας, περιμένω αυτή την έκθεση, προσβλέπω στην έκθεση που θα συστήσει μέτρα που θα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι δεν έχουν γίνει πολλά στον τομέα αυτό. Ίσως χρειάζεται μελέτες και άλλες συγκρίσεις, να δούμε τι γίνεται σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται όσον αφορά τους φόρους, τις συντάξεις, που όλα αυτά τα μέτρα ίσως επηρεάζουν τις γυναίκες σε κάθε χώρα διαφορετικά. Ευχαριστούμε την κυρία Μπράτνερτ. Το λόγο τώρα στην κυρία Αντρέα Σέσκοβα από τους Συντηρητικού στην Ευρώπη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, Madam President. And... Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρα. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στις μονογαμικές οικογένειες είναι η σημαντικότερη κατηγορία κατά την άποψή μου. Και αυτό σε συνάρτηση με τη φτώχεια και την πτυχή του φίλου στην φτώχεια. Θα ήθελα να δείξω ποια είναι η τσεχική άποψη, διότι κατάγομαι από τη Τσεχία, είναι η χώρα μου η Τσεχία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο 9% των Τσέχων μπαίνουν στη φτώχεια πέφτουν κάτω από το κατόφλιο της φτώχειας. Χαμηλό όριο, συγκρίνοντας με το μέσο όρο του 17% που είναι ευρωπαϊκός μέσο όρο. μέσος όρος. Τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν ότι η διαφορά μεταξύ φτωχών και πλουσίων στη χώρα μου είναι μικρότερη. Σε συγκρίση με τα άλλα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Παρ' όλα αυτά ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο τη φτώχεια. Οι πλέον ευάλωτε κοινωνικές ομάδες είναι παρόμοιες με αυτές που είναι και στα άλλα Αλλά για στις μονογονικές οικογένειες έχουμε μεγαλύτερη αύξηση στις μοναχικές μητέρες. Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό. 90% της ομάδας. Αυτή η ομάδα των ανθρώπων έχει το καλύτερο κίνδυνο για φτώχεια. Γιατί έχουμε γονείς χωρίς σύντροφο, με ένα μικρό παιδί, που να βρουν πλήρη απασχόληση πρέπει να λύσουν πολλά προβλήματα. Έλλειψη δουλειά, πρέπει να βρουν δουλειά με ευέλικτο ωράριο. Uh, Και δεν υπάρχουν ε, υπηρεσίες ε, για τα παιδιά που να τι επιτρέψει να δουλέψουν. Αυτό είναι βασικό πρόβλημα. Αυτοί οι μοναχοί γονεί προτιμούν να εργάζονται πιο πολύ ε, ε, σαν υπάλληλοι αλλά θα θέλαν να έχουν ευέλικτο ωράριο σαν υπάλληλοι. Ή θα προτιμούσαν μια δουλειά που θα μπορούν να δουλέψουν από το σπίτι του. Οι μοναχικέ μητέρε και οι πατέρε έχουν αυτό το πρόβλημα. Και οι πατεράδε. Είναι ευάλωτη η κοινωνική ομάδα. Και υπάρχουν λίγα προγράμματα στήριξή του. Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην απασχόληση και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Προγράμματα και εργαστήρια που βοηθούν τους μοναχικούς αυτούς γονείς να ενταχθούν στην αγορά εργασίας είναι καλά και που παρέχουν την αναγκαία δομή για μέρημνα των παιδιών. Είναι βασική ανάγκη αυτή. Θα βοηθούσε να λύσει το πρόβλημα της στόχιας αυτή η προσέγγιση. Πρέπει να αλλάξει η κοινωνική ευαισθητοποίηση όσον αφορά το πρόβλημα. Πρέπει να δουλέψουν σκληρά και τα άλλα και η Τσεχία για να τα βελτιώσουν αυτά. Προσβλέπω σε στενή συνεργασία στο μέλλον όσον αφορά το θέμα. Σας ευχαριστώ την προσοχή σας. Thank you. And... Τώρα ο λόγος στην κυρία Παβανόβα, σκιώδη εισηγήτρια, από τους φιλελεύθερους δημοκράτες της Ευρώπης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ήρθε τη σωστή στιγμή αυτή η έκθεση. Είναι πολύ δύσκολο θέμα αυτό, το θέμα της στόχιας. Δεν είναι μόνο θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορά τις γυναίκες, αλλά περνάμε οικονομική και χρηματοστητική κρίση. Και τώρα ξεκινήσαμε να συζητούμε και τη δημογραφική κρίση. Και χαίρομαι ιδιαίτερω που ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κ. Μπαρόσο, έθεσε σαν προτεραιότητα τη δημογραφική κρίση για την επόμενη δεκαετία. Και πιο πέρα θα είναι πρόβλημα. Αναφέρομαι στη φτώχεια λοιπόν. Συναρτήσει της δημογραφικής κρίσεως και στην έκθεσή σας θα βρείτε το σωστό σημείο να τονίσετε το θέμα αυτό. Υπάρχει μια ιστορική κληρονομιά όσον αφορά τη της γυναίκας στην κοινωνία. Όχι από οικονομική σκοπιά μόνο, αλλά και από κοινωνική. Πάνω από αυτό, με τη δημογραφική κρίση, επιδεινώθηκε η κατάσταση και είναι καλό να δούμε ποιες είναι οι τάσεις, οι αρνητικές τάσεις, οι οποίες συμβάλλουν σε αυτή την κακή κατάσταση. Υπάρχει και κάτι άλλο που θα πρέπει να εξετάσουμε εκ του σύνεγγυς. κυρίως με τις τελευταίες εκθέσεις που είδαμε για το εμπόριο ανθρώπων και τι γίνεται με τις γυναίκες από Τι έγινε πρόσφατα στη Γαλλία. Αυτό που έγινε ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε παρά να το προσέξουμε. Διότι είναι ένα πρόβλημα που συμβαίνει στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, αλλά τώρα αντιμετωπίζεται και από πολλές άλλες χώρες. Και δεν μπορούσαμε εμείς να ρίχνουμε τον μπαλάκι ένα στον άλλον από χώρα σε χώρα και να στείλουμε το πρόβλημα πίσω στη χώρα καταγωγής. Πρέπει να εξεταστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως, διότι είμαστε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Δεν είμαστε κλειστές κοινωνίες και ο καθένας φροντίζει τον εαυτό του. Γι' αυτό νομίζω ότι αν στην έκθεσή σας αναφέρετε συγκεκριμένα τις γυναίκες των μειονοτήτων, αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για όλους. Και ελπίζω ότι με αυτή την έκθεση και με τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής μας θα είμαστε σε θέση κάπως να προωθήσουμε την πρωτοβουλία της κυρίας Ρέντινγκ, της Επιτρόπου Ρέντινγκ, να καταλήξουμε σε αποτελεσματική στρατηγική για τις γυναίκες. Όσον αφορά την πρόταση παρουσίαση, εγώ δεν είδα να γίνονται πολλά. Ελπίζω να συμβάλλει η έκθεσή σα, ώστε να προωθηθεί το θέμα. Thanks, Mrs. Pavanova. Ευχαριστούμε την κυρία Παβανόβα. Τώρα θα δώσω, θα δώσω το λόγο στην κυρία Παρασκευά, που ασχολείται με τα θέματα τα κοινωνικά και τις πτυχές που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση και γενικότερα τις κοινωνικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο σε εσά, κυρία Παρασκευά. Παρακαλώ. Ε, thank Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ την Επιτροπή που μας ε, προσκάλεσε ούτω ώστε να μπορέσουμε να αντα... ανταλλάξουμε απόψεις στη δημόσια αυτή ακρόαση για τις γυναίκες και τη φτώχεια προσωπικά πριν την εξαετία μου στη μονάδα για τη φτώχεια είχα εργαστεί για 10 χρόνια στην μονάδα την υπεύθυνη για την ισότητα των φίλων και είμαι επιφορτισμένη ακόμα στο να εξετάζω τις πλέον ευάλωτες ομάδες γυναικών στα πλαίσια των εργασιών της μονάδας μου. Να αναφερθώ σε κάποια θέματα που εφήγησαν σήμερα. Και μετά, αν υπάρχουν ερωτήσεις, θα μπορούσα να απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, ξεκινώ από αυτό που η εκπρόσωπος του WAVE, η κυρία Webhofer, ανέφερε. Δηλαδή ότι η βία δεν συμπεριλαμβάνεται στη συζήτηση για τη φτώχεια. Και αυτό πάει και με το άλλο θέμα του εμπορίου ανθρώπων. Και αυτό λείπει από τη συζήτηση για τη φτώχεια. Προσπαθούσαμε σκληρά να πείσουμε τους συναδέλφους που είναι επιφορτισμένοι με αυτά τα θέματα σε άλλη γενική διεύθυνση να συμπεριλάβουν τη φτώχεια ανάμεσα στα αίτια εκείνα που μπορούν να οδηγήσουν στη βία και στο εμπόριο ανθρώπων. Και να τονίσουμε ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορούν να είναι συνέπειες αυτών των φαινομένων. Και είδαμε ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το οποίο υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ασχολείται κυρίως με τη βία και το εμπόριο γυναικών καλύπτει και αυτές τις πτυχές. Όμως, κατά το παρελθόν, στα πλαίσια της διαδικασίας κοινωνικής εντάξεως, εξετάζαμε αυτά τα φαινόμενα επίσης. Εδώ και κάποια χρόνια εστιαζόμαστε περισσότερο επί προτεραιοτήτων όπως είναι η φτώχεια των παιδιών και η ενεργός ένταξης αυτό δεν μας εμποδίζει όμως από το να εξετάσουμε και τη βία και το εμπόριο ανθρώπων. Το πρόγραμμα Oxfam, το οποίο αναφέρθηκε, χρηματοδοτήθηκε από το τμήμα μας για την κοινωνική ένταξη κοινωνική προστασία, για την εξίσωση των εισοδημάτων. Αυτό είναι μεγάλο θέμα στα νοικοκυριά, διότι ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζουμε τώρα το ποσοστό εισοδήματο στα νοικοκυριά δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική θέση των γυναικών. Και προβλέπεται ότι στα πλαίσια της νέας στρατηγικής για την ισότητα των φύλων για τα έτη 2010 μέχρι 2015, κάτι που υθετήθηκε μόλις τώρα, αυτό θα είναι κάτι που θα καλύπτεται, παρά το γεγονός αυτό όμως, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός των γυναικών αναφέρεται αόριστα στα πλαίσια του κεφαλαίου της οικονομικής ανεξαρτησίας. Βεβαίως, μεγαλύτερη προσοχή θα μπορούσε να δοθεί στο θέμα αυτό. Πράγματι, η φτώχεια πλήττει τις γυναίκες και στην Ανατολή και στη Δύση και με διαφορετικό τρόπο. Αλλά αυτό είναι και ένα θέμα μέτρησης. Πάντα χρησιμοποιούσαμε το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για να προσμετρήσουμε τη φτώχεια. Δηλαδή το 60% του μέσου εισοδήματο. Τώρα, σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρώπης για το 2020, πανέφερε η κυρία Ζήμερ, έχουμε άλλους δύο δείκτες για να κάνουμε τη μέτρηση. Στέρηση, ηλική στέρηση και τα άνεργα νοικοκυριά. Αυτά τα στοιχεία έχουν προσθεθεί στον υπολογισμό που κάνουμε για τα διάφορα κράτη-μέλη και αυτό βεβαίω θα θέσει και θέμα συγκρισιμότητα στοιχείων. Διότι τα κράτη-μέλη θα μπορούν να επιλέξουν ποιου ή μάλλον ποιον από τους τρεις δείκτε θα χρησιμοποιήσουν για να καταλήξουν στο στόχο τους. Να πετύχουν το στόχο που έχει καθοριστεί από τη στρατηγική την Ευρωπαϊκή το 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ποιες είναι οι πλέον ευάλωτες ομάδες γυναικών και επικεντρώνει τις προσπάθειές της επί των νεωτέρων γυναικών που θέλουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, επί των ηλικιωμένων γυναικών και των συνταξιούχων και βεβαίως των ε, μητέρων μέλη, που είναι μέλη μονογαμικής, ε, μονογονικής οικογένειας. Και τέλος, έχει γίνει κάποια προσπάθεια, έχει ξεκινήσει η προσπάθεια εδώ και 15 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τον εντοπισμό των δικαιωμάτων όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ενδεχομένω θα μπορούσε να προωθηθεί κυρίως διότι θα μπορούσε να συνδέεται με όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται ούτως ώστε να επιτευχθεί η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών. Αυτά από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ώρα. Θα μπορέσω να απαντήσω ενδεχομένω ερωτήσει αργότερα και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα φτάσαμε στι ερωτήσεις. Η κυρία Λούνατσεκ θέλει πρώτα. Και παρακαλώ να είσαστε σύντομοι. Thank you Um... Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών και την Επιτροπή Γυναικών που ε, οργάνωσε αυτό το πάνελ και συμπεριέλαβα και το θέμα της βίας. Δεν το λέω εδώ γιατί είναι η κυρία Βίπ Χόφερ και είναι από την ίδια χώρα, είναι συμπατριώτησά μου. Και εγώ εδώ και 30 χρόνια προσπάθησα να δημιουργήσω το πρώτο καταφύγιο γυναικών στο Τιρόλο, πολύ συντηρητική περιοχή της Αυστρίας. Ξέρω τι σημαίνει κάτι τέτοιο αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτή η διάσταση της βίας να συμπεριληφθεί στο θέμα της στόχιας. Και η κυρία Βεπχόφερ άριστα το έκανε αυτό, αναφερόμενη στο ζήτημα εφορά την υγεία, την παιδεία, την απασχόληση. Είναι κάτι που επηρεάζει τις γυναίκες περισσότερο από ό,τι οι άντρες. Η βία κατά των γυναικών σε όλα τα επίπεδα. Και όταν μιλάμε συχνά για τη φτώχεια, οι γυναίκες κερδίζουν λιγότερα, έχουν λιγότερη επιρροή στη λήψη αποφάσεων οι γυναίκες, αυτό το ξέρουμε όλοι. Όμως, περίληψη της βίας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι είναι κάτι αόρατο πολύ συχνά, δεν υπάρχει ο συσχετισμός και είναι κάτι που μοιάζει με τη φτώχεια. Σχετίζεται με την τροπή, το όνειδος, κάτι που δεν θέλει κανείς να αναφέρει η ντροπή είναι κάτι το οποίο δεν θα το συζητούν οι γυναίκες. Μάθαμε να το συζητούμε, ήταν δύσκολο για τις περισσότερες, αλλά είναι κάτι που ακόμα δεν φαίνεται. Η φτώχεια είναι κάτι παρόμοιο. Δεν θέλει κανείς να μιλάει για τη φτώχεια του. Θέλει να δείξει ότι μπορεί να αγοράσει κάτι για τα παιδιά του, για τον εαυτό του, ότι έχει ε, φορά καλά ρούχα. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτές οι δύο πτυχές της φτώχεια και της βίας να ενταχθούν και να δούμε πώς αυτά οδηγούν στη φτώχεια και να συμπεριφθούν στην έκθεση. Και το άλλο θέμα που αναφέρθηκε των ατομικών δικαιωμάτων, της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών, να έχει το δικαίωμα να πάρει σύνταξη όταν γεράσει, να μην εξαρτάται από ένα σύζυγο που μπορεί να έχει ή να μην έχει στο μέλλον ή πόσα χρήματα κερδίζει ο σύζυγος και όχι η ίδια γυναίκα. Τα συνταξιωτικά συστήματα θα πρέπει να γίνουν ε, τέτοια, ώστε να, να διεκδικεί η γυναίκα τα δικαιώματά της, είτε είχε διαβίου ε, δουλειά ή όχι. Ε, να υπάρχουν νόμοι που λέει μικρά ποσά μπορεί να καταβάλει κάθε μία μετά τα 18 και να έχει δικαίωμα συνταξιοδότηση όταν γεράσει. Και τα ατομικά δικαιώματα για τι μετανάστριες. Αναφέρθηκε αυτό. Θα ήθελα να ξέρω ίσω και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να μπει στην έκθεση. Υπάρχει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, δίνει το δικαίωμα στη μετανάστρια που ήρθε, παντρεύτηκε και έχει δικαίωμα διαμονή μόνο επειδή παντρεύτηκε μετανάστη ή ηθαγενή, γηγενή και πάρει διαζύγιο, έχει δικαίωμα να μείνει τα μόνη τη. Στη Γερμανία, στη χώρα μου, στην Αυστρία, δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Σε χώρε δεν ξέρω τι γίνεται. Θα ήταν ενδιαφέρον και αυτό να αναφέρεται στην έκθεση, να δούμε τι γίνεται. Ποιε χώρε το προβλέπουν αυτό, το υποστηρίζουν και να ζητήσουμε και τι άλλε να κάνουν το ίδιο. Και στο τέλο, για μια τέτοια έκθεση τι πρέπει να δούμε. Είχαμε 30-40 χρόνια το φεμινιστικό κίνημα που θέλαμε να γίνουν κάποια πράγματα, αλλά εξακολουθούμε να ζούμε σε πατριαρχικές δομές. Άρα είναι σημαντικό ως πολιτικοί που έχουμε γίνει, εμείς που είμαστε εδώ στο Κοινοβούλιο, να έχουμε μια έκθεση που όπως προαναφέρθηκε σπρώχνει, πιέζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την πιέζει να προχωρήσει και την κυρία Ρέντινγκ να τους πρόξουμε ώστε να κάνουν κάτι αποτελεσματικό, διότι τόσα πράγματα συζητήσαμε τόσο μακρόν δράση, ε, σχέδια δράσης. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν του νόμου και τι δράσει και όλα αυτά να υλοποιηθούν σε, σε πράξεις. Uh, Η κυρία τώρα θα πάρει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Υπάρχουν δύο σχόλια ή μάλλον ερωτήσεις που θα ήθελα να κάνω. Συζητήσαμε για το πόσο με... πολλές είναι πόσο πολύ πλήττονται οι μονογονεϊκές οικογένειες από τη φτώχεια. Επίσης, ε, υπόθηκε ότι είναι πολύ σημαντικό να αξιολογήσουμε τη δημογραφική διάσταση και θα ήθελα να το τονίσω. Βλέποντας την έκθεση που εκπονήσατε, ε, κυρία Πλάμ, μας βλέπουμε ότι τα οικονομικά επιχειρήματα θα πρέπει να είναι πολύ πιο ξεκάθαρα, γιατί αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε πείνα σε πολλές χώρες, όπως είναι για παράδειγμα η Βουλγαρία. Και αυτοί που προέρχονται από μειονότητες με πολύ χαμηλές αποδοχές, όπου ο αριθμός των παιδιών είναι ιδιαίτερος υψηλός, πολύ συχνά τα παιδιά αυτά αποκλείονται από την κοινωνία, δεν έχουν πρόσβαση στην παιδεία, δεν έχουν, δεν έχουν σωστές παροχές ε, περίθαλψη Και η κατάσταση είναι ιδιαίτερο δεινή. Είναι πολύ σημαντικό να δοθεί έμφαση ότι στην παρούσα συγκυρία σε πολλές ε, χώρες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης διακυβεύεται ίδια τους η αξιοπιστία εάν ε, συνεχίσουν να παραμελούν τους γονείς ή τα παιδιά εκείνα που αναπαράγουν ακριβώς αυτές τις καταστάσεις ένδυες και φτώχες. Θα πρέπει λοιπόν να στρέψουμε εδώ την προσοχή μας. Θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας πλέον. Γιατί αυτή τη στιγμή άλλαξε το σύστημα στην Ανατολική Ευρώπη και οι άνδρες που χάνουν τις θέσεις εργασίας, που δημιουργούν τέτοια ένταση εντός της οικογένειας, όπου πλέον οι ρόλοι έχουν αλλάξει ριζικά και η κυριαρχία του άνδρα υπό την οικονομική έννοια έχει αλλάξει πλέον ακόμα και εκεί. Και αυτό βάζει τη γυναίκα σε εντελώς διαφορετική κατάσταση. Υπάρχει μια μεγάλη ποσότητα ψυχικού άγχους που δεν μπορούν να αντέξουν οι άνθρωποι αυτοί, οι γυναίκες αυτές, προσπαθώντας να θρέψουν σωστά τα παιδιά τους και να έχουν και μία θέση στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε έγκαιρα. Ε, νομίζω ότι οι δείκτες μπορούν να μας προσφέρουν κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία εν σχέση με τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι οικογένειες. Και δεν έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει όλα να τεθούν υπό την ε, προοπτική του φύλου. Αλλά θα πρέπει να μιλάμε για τι γενικέ αυτέ σαν άτομα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασία, ζουν μακριά από τα αστικά κέντρα, είναι άνεργε, δεν έχουν δημόσια υπηρεσίε, έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, ε, έχουν κοινωνικέ εντάσει, υφίστανται κοινωνικέ διακρίσει κλπ. Είναι ένα ολόκληρο πλέγμα εθνοτική συχνά φτώχεια, η οποία αναπτύσσεται Ω ως κοινωνικό φαινόμενο και αναπαράγεται σε αυτά τα στρώματα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αποστείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σχέση ακριβώς με το οικονομικό επιχείρημα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γερόκα και τώρα θα δώσω το λόγο στους ε, ομιλήτριες για να σχολιάσουν. concerning the questions we have got from our colleagues. And first of all... Λοιπόν, θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Βεπχόφερ. Και παρακαλώ προσπαθήστε να είστε σύντομοι γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μας. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε αυτή τη σχέση μεταξύ βίας και κατά των γυναικών και φτώχειας. και ε, στην έκθεσή μου φωτίζονται αυτές οι διασυνθέσεις. Σας περίγραψα πώς είναι η κατάσταση στην Αυστρία. Νομίζω ότι μπορούμε να αναμένουμε σημαντικές βελτιώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να δούμε τη θέση των μεταναστριών, των ε, γυναικών με ειδικέ ε, ανάγκες κλπ. Κάτω από αυτό το πρίσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Πόπ. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε εδώ. Θα ήθελα να πω να τονίσω την κατάσταση μιας γυναίκας σε μονονογική οικογένεια που έχει ένα παιδί με ειδικέ ανάγκες, για παράδειγμα. Ε, παιδί που χρειάζεται μια συνεχή φροντίδα και σχέση με τις παρατηρήσεις που, έκανε, που έκαναν συνάδελφοι από την Αυστρία, θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή οδηγία του 2004 που δεν επιτρέπει στις αρχές να αρνηθούν το δικαίωμα διαμονής στη μετανάστρια γυναίκα με το επιχείρημα ότι έχει διαζευθεί κλπ. Θα ήταν κατάχρηση υπό την έννοια τη οδηγία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. My mother tongue. Και τώρα θα προσπαθήσω να μιλήσω στη δική μου γλώσσα. Ευχαριστώ τις καλεσμένους μας επίσης τις συναδέλφισες για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και θα συνεχίσουμε στο επόμενο θέμα που έχουμε σήμερα σε διάταξη, το οποίο είναι η, η γενικότερη στόχη για τη μείωση της φτώχειας και ποιες, ποια είναι τα μέτρα και ποιες οι καλύτερες πρακτικές. Λοιπόν, αν τώρα οι καλεσμένες ε, ε, οι εμπειρογνώμονες που έχουμε καλέσει θα ήταν καλό να έρθουν εδώ στο ε, Προεδρείο. Να ευχαριστήσω όμως τις, το, το προηγούμενο πάνελ. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ για τη συμμετοχή στη συζήτηση αυτή. Παρακαλώ. Λοιπόν, καλωσορίζω τους καλεσμένους μας στο δεύτερο μέλος της συζήτησης που αφορά τους γενικότερους στόχους για τη μείωση της φτώχειας και ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές. Χαίρομαι λοιπόν που καλωσορίζω εδώ σήμερα την Anne-Sophie Parents που είναι διευθύντρια της AGE, μια, ένας οργανισμός ομπρέλα για θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για των ηλικιωμένων. Καλώ ήρθατε λοιπόν σε αυτήν εδώ την ακρόαση και θα πάρετε αμέσως το λόγο. Παρακαλώ. Thank you very much and, uh, thank... Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πράγματι, εδώ μιλάω εκ μέρους του AIDS, Ευρωπαϊκού Δικτύου που αντιπροσωπεύει 156 οργανώσεις μέλη, 28 εκατομμύρια ηλικιωμένου συναθρίζουμε, οι περισσότερες είναι γυναίκες όπως τα φαντάζεστε. Ε, ήμουνα πρόεδρο της κοινωνικής πλατφόρμας, δεν είμαι πια, αλλά βέβαια ακόμα το θέμα της ηλικία είναι θέμα της κοινωνικής πλατφόρμας. Μου ζητήθηκε να αναφερθώ ακροθυγώς στο ειδικό κίνδυνο της φτώχειας που αντιμετωπίζουν ηλικιωμένες γυναίκε όταν φτάσουν την ηλικία συνταξιοδότησης. Για μα πράγματι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα, κρισίμου σημασία ζήτημα, Κυρίω στα σημερινά πλαίσια, διότι όπω ξέρετε αντιμετωπίζουμε οικονομική κρίση. Και ξέρουμε ότι γίνονται σημαντικέ μεταρρυθμίσεις, ριζικέ, και ανησυχούμε τα μάλα, διότι αυτέ οι μεταρρυθμίσεις εισάγονται χωρίς να εξετάζεται επαρκώς η διάσταση των φύλων και τι συνέπειες θα έχει αυτό για τις ηλικιωμένες γυναίκες πιο συγκεκριμένα. Το ξέραμε και πριν από την κρίση ότι οι ηλικιωμένε γυναίκε και άντρε υπέφεραν από ανισότητε όσον αφορά την κοινωνική προστασία. Οι ηλικιωμένε γυναίκε έχουν μικρότερη πρόσβαση στην επαρκή κοινωνική προστασία, κυρίω όσον αφορά τα συνταξιδοτικά ζητήματα. Επίση, υπήρξε και διάκριση όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη όσον αφορά τι γυναίκε ηλικιωμένε. Ο τομέα των συντάξεων είναι ο βασικό τομέα και συνδέεται άρρηκτα αυτό με το εισόδημα και την ικανότητα να ζήσει κανείς αξιοπρεπή ζωή σε, όταν είναι σε μεγάλη ηλικία. Γίνεται εδώ των γυναικών, πρώτα απ' όλα επειδή είναι γυναίκες, αναφέρθηκε αυτό, αλλά και λόγω της ιστορίας γονιμότητας δεν έχουν επαρκή αποζημίωση για ε, τις διακοπές καριέρας. Έχουν συντομότερες καριέρες οι γυναίκες ε, από ότι άντρες και πιο σύντομες καριέρες για να έχουν τη σωστή σύνταξη. Αυτό δεν καλύπτεται από τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται. Αντίθετα, παρατείνουμε την ηλική εργασία, το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι χρειάζεται για να υπάρχει η βιωσιμότητα της κοινωνικής προστασίας. Αλλά δεν αποζημιώνεται επαρκώς η διακοπή καριέρας που κάνει η γυναίκα. Και δικαιολογημένε διακοπέ. Και αυτό επηρεάζει αυτέ που έχουν χαμηλό εισόδημα, που δεν έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύσουν κάποια χρήματα, να έχουν και κάποια χρήματα στην άκρη πέρα από τι ξέρουμε ότι υπάρχει και μια τάση που αυξάνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να απομακρυνόμεθα από τις δημόσιες συντάξεις του πρώτου πυλώνα, που εξορισμού είναι, πώς να το πω, πιο αλληλέγγυες και έχω μηχανισμό που αποζημιώνει εκείνους που παίρνουν πολύ χαμηλή σύνταξη και μπορούν να έχουν πικουρική σύνταξη. Όταν φύγεις από τα δημόσια αυτά σχήματα, πας στον ιδιωτικό τομέα. Εκεί, δυστυχώς, οι γυναίκες δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα σε σχέση με τους άντρες. Κάποιος, αν έχει δικό του συνταξιωτικό ταμείο, είναι εργοδότης, λέει ναι, αλλά οι γυναίκες ζουν περισσότερο. Οπότε τελικά παίρνουν περισσότερα. Αλλά έχουν το ίδιο ποσό για να ζήσουν πιο πολλά χρόνια. Πρώτα απ' όλα βέβαια δεν παίρνουν τα ίδια ποσά, διότι πολλές γυναίκες εργάζονται το μίσο που δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτές τις συντάξεις που δίνουν αυτοί οι εργοδότες συγκεκριμένοι και μετά πρέπει να αγοράσει κανείς ιδιωτική ασφάλιση. Οπότε υπάρχει διάκριση εναντίον της γυναίκας. Διότι οι εταιρείε βασίζουν τους υπολογισμούς σε παλαιούς πίνακες μακροζωίας για τις γυναίκες που βασίζονται στη μακροζωία των γυναικών που δεν έχουν εργαστεί πολύ. Άρα για την ώρα έχουμε μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες. Αλλά υπάρχουν κάποιες προβολές και υπολογισμοί που δείχνουν ότι το προσδόκιμο ζωής των γυναικών θα πλησιάσει πολύ των ανδρών. Για τις εργαζόμενες γυναίκες θα πλησιάσει το προσδόκιμο ζωής των ανδρών. Γιατί, γιατί είναι η ζωή μας πάρα πολύ δύσκολη. Μπορεί να μας βοηθάνε οι ορμόνες, αλλά τις καταναλώνουμε τις ορμόνες, διότι έχουμε διπλό βάρος όταν εργαζόμαστε έχουν περισσότερο στρες, περισσότερα προβλήματα υγείας. Πέραν λοιπόν αυτού, δηλαδή ότι φεύγουμε από τις δημόσια χρηματοδοτούμενες συντάξεις, υπάρχει ένα άλλο θέμα που συζητά το Κοινοβούλιο. Η αναθεώρηση του άρθρου 5 της Οδηγίας για την Ισότητα των Φύλων. Μέσω του λόμπινγκ των κρατών μελών και της βιομηχανίας του τομέα συμφώνησαν τα συντηρητικά ταμεία να κάνουν διακρίσεις βάσει του φύλου. Άρα υπάρχει ένα ποσό σύνταξης, αλλά επί μήνες το κέρδος, το επιτόκιο επενδύσεως από αυτό το ποσό είναι πολύ χαμηλότερο. Το κόστος της ζωής είναι το ίδιο. Μπορεί η γυναίκα να ζει κάποια χρόνια παραπάνω, αλλά τα χρήματα που χρειάζεται το μήνα είναι τα ίδια. Και αυτό προσπαθούμε να το καταπολεμήσουμε. Ποιε είναι οι λύσει, λοιπόν. Πολεμάμε ούτω ώστε να απαλλαγούμε από αυτή τη διάκριση των συνταξιδοτικών ταμείων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που επιτρέπεται να κάνουν λόγω των φίλων. Θέλουμε να υπάρχει ενίως unisex πίνακας. Να πούμε στα κράτη-μέλη, αν φεύγετε από τα δημόσια συστήματα, τα συνταξιδοτικά που είναι αλληλέγγυα και πάτε προς τα ιδιωτικά συνταξιωτικά ταμεία, θα πρέπει να εξασφαλίσετε ταυτόχρονα ότι εφαρμόζετε κατάλληλα μέτρα, τόσο ώστε οι γυναίκε να μην υποφέρουν από αυτή τη μετακίνηση. Ότι θα αντιμετωπιστούν ισότιμα όσον αφορά τα αποτελέσματα, όχι όσον αφορά το ποσό που, που, που βάζουν στην άκρη. Διότι βγάζει μια γυναίκα 15% λιγότερο στην ίδια θέση εργασία με τι ίδιε δεξιότητε. Άρα έχουμε λιγότερα χρήματα να βάλουμε στο ιδιωτικό συνταξιωτικό ταμείο και ταυτόχρονα τα ιδρύματα δίνουν λιγότερα κέρδη για τα χρήματα που επενδύουμε. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να αυξηθεί η φτώχεια τα επόμενα 20-30 χρόνια σε ηλικιωμένες γυναίκες. Θέλουμε λοιπόν να εισαχθεί προσδόκιμο, πίνακες προσδοκίμου ζωής, θνησιμότητας που θα είναι unisex, ίδια οι συντελεστέ για άντρε και γυναίκε. Και όταν τα κράτη-μέλη φεύγουν από τα κρατικά συστήματα ή πάνε στα ιδιωτικά, δεν το συστήνουμε αυτό, αλλά αν οι πολίτε το θέλουν στο κάτω-κάτω, λέμε άμα γίνει αυτή η αλλαγή θα πρέπει να εξασφαλίζουν τουλάχιστον εκείνα τα συστήματα θα είναι υποχρεωτικά και ότι θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνο που ξοδεύει η γυναίκα για να προσέχει του ηλικιωμένου, να μεγαλώνει παιδιά ή ε, να βοηθά κάποιου συγγενεί και διακοπές καριέρας. Ε, θα πρέπει να είναι αλληλέγγυο το σύστημα. Υπάρχουν κάποια ιδιωτικά τέτοια σχήματα τα οποία είναι αλληλέγγυα και τα οποία δίνουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Θέλουμε επίσης πρώτα απ' όλα να καταπολεμήσουμε την έλλειψη επάρκειας συντάξεων καταπολεμώντας τη διάκριση τις οποίες είναι θύματα οι γυναίκες στην αγορά εργασίας. Μειώνοντας τις διαφορές σοφά την καριέρα και τις αμοιβέ, αυτή είναι η αφετηρία, Θέλουμε η στρατηγική της Ευρώπης του 2020 να εισαγάγει μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν τη συμφωλίωση οικογενειακής ζωής και φροντίδας με τον επαγγελματικό βίο. Αυτό επανειλημμένα έχει υποθεί γιατί το τονίζουμε εκ νέου, διότι παρατηρούμε ότι αυτό είναι ένας τομέας στον οποίο η τοπική αυτοδίκηση αντιμετωπίζει σοβαρές περικοπές και περικόπτονται οι διαθέσιμες υπηρεσίες. Άμα περικόψεις τη υπηρεσία περίθαλψης, ποιοι υποφέρουν ξανά οι γυναίκες διότι η φροντίδα των ηλικιωμένων θα πέσει ξανά πάνω τους. Αυτό σημαίνει ότι για τους 45 συν οι γυναίκες περισσότερο θα πρέπει να αποσύρονται από την αγορά εργασία και να πάρουν μερική απασχόληση για να φροντίσουν τους εξαρτώμενους ηλικιωμένου. Και αυτό θα έχει συνέπεια στα δικά τους συνταξιδοτικά δικαιώματα. Λέμε επίσης ότι το θέμα της ε, συντάξεως εκείνων που επιβιώνουν είναι κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Οι χείρες πολλές χείρες πρέπει να ζήσουν με τη σύνταξη που παίρνουν από την ε, σύνταξη του Μακαρίτη. Επίσης, είναι ανεπαρκή πολύ συχνά οι συντάξει και δεν παίρνουν ατομικά δικαιώματα. Κάποιες γυναίκες υποχρεώνονται να μείνουν με το σύζυγό τους γιατί διαφορετικά μένουν χωρίς κάποιο εισόδημα όταν φτάσουν στην ηλικία συνταξιοδότηση. Θέλουμε και καλύτερες εικόνες να διαμορφωθούν μέσω του ΟΣΑ, των Ερευνητικών Ιδρυμάτων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ούτω ώστε αυτοί που διαμορφώνουν πολιτική να μπορούν να αξιολογούν καλύτερα τι συνέπειε έχουν οι μεταρρυθμίσει επί τέτοιων ομάδων όπω είναι οι γυναίκε. Διότι για την ώρα χρησιμοποιούν πίνακε που βασίζονται σε εικόνα, που βασίζονται σε άντρα που βγάζει τα χρήματα και απασχολείται πλήρω. Και μεταρρυθμίσει που εισάγουν βλέπουν πώ επηρεάζουν αυτό το προφίλ. Και ξέρουμε βέβαια ότι οι συντάξεις θα έχουν μειωθεί, αλλά προχωράνε στο βαθμό που θεωρούν δυνατόν ούτω ώστε να επανεκλεγούν και να παραμείνουν δημοφιλείς οι πολιτικοί. Αυτό το προφίλ που χρησιμοποιούν δεν ταιριάζει με τις ανάγκες των γυναικών και σίγουρα πολλών ανδρών που έχουν συντομότερες καριέρες. Εάν μειώνονται σημαντικά οι συντάξει, καμιά φορά μέχρι 40% σε κάποιε χώρε. Είναι 40% σε σχέση με το μισθό που έπαιρνε πριν τη σύνταξη. Αν μειωθεί τόσο το εισόδημα, ε, θα είναι πιο μεγάλη η διαφορά για τις γυναίκες. Γίνεται σχετισμός μεταξύ εισφορών μεγαλύτερος τώρα και συντάξεις που χορηγείται. Και όσο μεγαλύτερη σχέση μεταξύ εισφορών και τελικής συντάξεως, τόσο πιο επώδυνο θα είναι αυτό για τις γυναίκες που εκτελούν και άλλα καθήκοντα πέτσι καριέρας. Εάν δεν μπορείς να δημιουργήσεις επαρκή στα δικαιώματα και δεν λαμβάνονται υπόψη οι διακοπές της καριέρας σου που, που παίρνεις για να φροντίσεις κάποιους, τότε θα αυξηθεί η διαφορά ανδρών γυναικών στη σύνταξη. Θέλουμε λοιπόν αυτή η εικόνα να βελτιωθεί, να γίνει έρευνα, εργαλεία να διαμορφωθούν για να αναπτύξουμε καλάθια καταναλωτών για του ηλικιωμένου, όπω τα αποκαλούμε. Να βάλουμε υπόψη το ότι όταν γερνάει κανεί, η σύνταξή του πολύ συχνά δεν ε, προσαρμόζεται κατάλληλα. Έχει πολύ πιο χαμηλή, ε, πιο χαμηλή σύνταξη από τη μια και από την άλλη αυξάνεται το κόστος για την πρόνοια, για, για τη φροντίδα που χρειάζεσαι. Θέλουμε αυτό το καλάθι να λαμβάνει υπόψη πραγματικέ ανάγκε των ηλικιωμένων και ιδιαίτερα των πολύ ηλικιωμένων. Τι χρειάζεται για να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή. Και αυτό το καλάθι μπορεί να το γεμίσει κανείς μέσω οικονομικής συνεισφοράς από τη σύνταξή τους ή και με άλλου τρόπους, όπως η είδος συνεισφορά. Αυτό γινόταν αρκετά. Ελεύθερες δημόσιες μεταφορές, ελεύθερη περίθαλψη υγειονομική, υποστήριξη για λογαριασμό στέγασης ή θέρμανσης. Αυτές είναι οι υπηρεσίες ή εισφορές εις είδος που έχουν περικοπεί λόγω της κρίσης που περνάμε. Χωρίς αύξηση της σύνταξης, αντιθέτως. Τελικό αποτέλεσμα είναι καταστροφικό, όπως καταλαβαίνετε, για τις γυναίκες με χαμηλό εισόδημα. Και δεν ξέρουν τι, να... δεν ξέρουν τι κάνουν τώρα. Ή μάλλον δεν θέλουν να δημοσιευθεί, να δημοσιοποιηθεί αυτό που κάνουν οι πολιτικοί. Θέλουμε εργαλεία να γίνει αξιολόγηση. Τι χρειάζεται κανεί να ζήσει αξιοπρεπώ. Είτε παίρνει αυτά που χρειάζεται από τη σύνταξή σου και μόνο. Ή όπω σε κάποιε χώρε χρειάζεσαι να αγοράσει συμπληρωματική επικουρική ασφάλιση για να μπορεί να συνεχίσει να καλύπτεσαι όσον αφορά την υγεία, γιατί αυτή είναι άλλη μια τάση που αντιμετωπίζεται. Βλέπουμε σε διάφορε χώρε ότι συμβαίνει αυτό και δημιουργούνται προβλήματα, διότι όσο πιο ηλικιωμένο είναι κανεί, τόσο πιο μεγάλο κίνδυνο για την ασφαλιστική εταιρεία, τόσο πιο δαπανηρή είναι η επικουρική ασφάλιση που θε να αγοράσει. Αποτέλεσμα, πάρα πολλοί ηλικιωμένοι, πολλοί ηλικιωμένοι χρειάζονται περίθαλψη και δεν ε, έχουν τα χρήματα να αγοράσουν την επικουρική ασφάλιση. Και πρέπει να περιμένουν μέχρι ώστε να αρρωστήσουν τόσο σοβαρά, τόσο ώστε να εισαχθούν στο νοσοκομείο. Και τότε αυτό είναι πιο δαπανηρό για την κοινωνία. Αυτά είναι τα λίγα στοιχεία, λίγε συστάσει που θα θέλαμε να κάνουμε. Κάνουμε εκστρατεία γι' αυτό. Μαζί ε, με άλλου φορεί προσπαθούμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση όσον αφορά αυτές τις διαστάσεις που αφορούν τις γυναίκες όσον αφορά τι συνταξιδοτικέ μεταρρυθμίσει και όσον αφορά τα συστήματα προνοία και τις μεταρρυθμίσεις τους. Χαιρόμαστε που η Βελική Προεδρία το θέμα αυτό το πήρε πολύ στα σοβαρά και ελπίζουμε ότι κάτι καλό θα βγει από αυτό, ε, κυρίως τα, συμβούλια του, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στο τέλος του έτους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις ενδιαφέρουσες ε, απόψεις στην εισήγησή σας και να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Άρτο Κόκχο, που είναι σύμβουλος στο Υπουργείο για τις Κοινωνικές Υποθέσεις στη Φιλανδία, στο τμήμα προγραμματισμού. Γεια σας, καλώς ορίσατε στην ε, δημόσια αυτή ακοράση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, λέει σας ειδικά ο κλασμένος. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση Φαίνεται ότι είμαι ο μόνος άνδρας εδώ, το μόνο σενικό. Εδώ στην... στους ομιλητές. Και αυτό μου θυμίζει μια... κάτι στην ιστορία. Το 2000, μια συνδιάσκεψη στην Πορτογαλία όπου ήταν ε, ένα συνέδριο στην διάσκεψη για την ισότητα των φύλων και υπήρξε μια τεράστια φιλανδική αντιπροσωπεία με νέα μέλη. Και εγώ ήμουν ο μόνος άνδρας σε αυτή την ομάδα. Ε, ίσως ε, είμαι τυχερός που μου συμβαίνει αυτό για δεύτερη φορά. Ε, θα ήθελα... Ε, η δική μου παρουσίαση είναι πιο θεωρητική ή τουλάχιστον αυτή την οποία είχα προετοιμάσει και δεν θα την ε, παρουσιάσω εδώ λεπτομεριακά. Θα ήθελα απλώς να περισσώ σε κάποια σχόλια. Έχω τέσσερα θέματα κατά νου. Και τα σχόλιά μου σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020. Ε, είμαι μέλος της Κοινωνικής Επιτροπής και για το λόγο αυτό ασχολούμαι με το προπαρασκευαστικό έργο στην ε, Φιλανδία για την διαδικασία αυτή και τα τέσσερα σχόλια που θα σας κάνω ε, βασίζονται ακριβώς ή απορρέουν μάλλον από την φιλανδική εμπειρία. Το πρώτο αφορά την οικονομική ύφεση. Και εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Η οικονομική ύφεση ενδεχομένως έχει μακροπρόθεσμες κοινωνικές επιπτώσεις. Αυτό το ζήσαμε στη Φιλανδία επίσης τη δεκαετία του 90, όπου είχαμε μια πολύ βαθιά ύφεση. Μακροχρόνιες λοιπόν κοινωνικές επιπτώσεις που μπορούν να παραμείνουν ένα βαρύ φορτίο για τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά συστήματα. Η ύφεση στη Φιλανδία τη δεκαετία του 1990 έδειξε ότι η μακροπρόθεσμη και διαρθρωτική ανεργία είναι τεράστιος κίνδυνο και δεν μπορεί, τεράστιο πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τα συνήθη κοινωνικά μέτρα. Και αυτή ήταν μια βασική εμπειρία που εντελήσαμε από την περίοδο της ύφεση. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχουν αριθμοί, στοιχεία μιας τεράστιας ανεργίας και θα είναι τεράστιες μακροπρόθεσμες ζημίες για τα, τις οικονομίες των χωρών μελών τα προσεχή χρόνια. Ε, ίσως τα πράγματα πάνε κάπως καλύτερα, αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να ζημιώσει τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας στις χώρες μέλη. Στη Φιλανδία είναι κυρίως ένα πρόβλημα για τους άνδρες αλλά μέσω άλλων μελών της οικογένειας και των παιδιών το πρόβλημα αυτό καθίσταται κοινό εντός του κοινωνικού συστήματος. Κατά δεύτερο λόγο, θα ήθελα να πω ότι η Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 θέτει προκλήσεις προς μια πολιτική που προσπαθεί να ευεργετηθεί από ποσοτικούς ε, στόχους. Στη Φινλανδία χρησιμοποίησαμε κοινωνικούς δείκτες και τους χρησιμοποίησαμε σε τακτά χρονικά διαστήματα και πολύ εκτεταμένα αλλά δεν έχουμε μια τέτοια παράδοση ποσοτικών δικτών. Έχουμε μόνο ένα πολιτικό πρόγραμμα αυτού του τύπου να μειωθεί ο αριθμός των αστέγων εντός μιας ε, κυβερνητικής θητείας. Στο κοινωνικό τομέα δεν έχουμε άλλα τέτοια παραδείγματα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι η παράδοση αυτή είναι αρκετά ασθενής στη χώρα μας. Και αυτό ισχύει και για άλλες χώρες μέλη, όπου είδαν το φως κάποια προγράμματα, αλλά όχι με τέτοιου είδους ε, στόχους ε, που να εκφράζονται σε αριθμούς. Έχουμε χρησιμοποιήσει κάποιους δείκτες και συστήματα παρακολούθησης για πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, αναθεωρήσαμε τον αριθμό των αποδεκτών ε, κοινωνικής ε, βοήθειας και την ε, εξέλιξη των αριθμών αυτών. Αλλά η πολιτική στοχοθεσία σε αριθμούς είναι μια εξαιρετικά δύσκολη δραστηριότητα. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, συνειδητοποιώντας ότι τα σχετικά μέτρα είναι δύσκολα, γιατί η αξιοπιστία μπορεί να οικοδομηθεί μέσω της διάδοσης, μέσω της ενημέρωσης και της βελτίωσης του επίπεδου αποδοχών. Η Γκαμπριέλ Τσίμερ ε, προηγουμένως σχολίασε σχετικά και είπε ότι τα 10 εκατομμύρια είναι υπερβολικά χαμηλός αριθμός και στη συνέχεια είπε ότι υπάρχει δυνατότητα για τις χώρες μέλη να επιλέξουν τους δικούς τους δείκτες. Βεβαίως το σχόλιο αυτό είναι σημαντικό, αλλά θα ήθελα να, πάω κάτι, να πω κάτι που πηγαίνει προς αντίθετη κατεύθυνση. Είναι σημαντικό η στοχοθεσία αυτή να γίνει και υπάρχει μια δυσκολία εδώ γιατί έχουμε να κάνουμε με αριθμούς και ιδιαίτερα όσον αφορά ε, αριθμούς σε για τις αποδοχές. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση, ωστόσο, να εργαστούμε και με αυτούς τους ε, δείκτες, προσπαθώντας να κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερα τη δουλειά μας. Δεν θα πρέπει να βασόμαστε μόνο στους αριθμούς, αλλά είναι πολύ σημαντικό να χαράξουμε μια σωστή τάση. Ίσως, ε, μα μακροπρόθεσμα θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να εμποδίσουμε την μείωση των αποδοχών με ποιοτικού όρους. Τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, κατά τρίτο λόγο, και οι δημόσιες υπηρεσίες είναι σημαντικές για τις οικογένειες με χαμηλές αποδοχές. Ε, και εδώ υπάρχει μια έντονη διάσταση φύλου. Μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι, για παράδειγμα, σε μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά ισχύει κάτι τέτοιο. Επιπλέον, οι σωστές ε, παροχές υπηρεσιών σχετίζονται με ανάγκες του κύκλου ζωής. Ε, τα δημογραφικά στοιχεία μας δείχνουν τι γίνεται με τους ολικιωμένους και πώς αυξάνονται αυτές οι ανάγκες. Αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η χάραξη σφαιρικών πολιτικών είναι σημαντικό στοιχείο για την καταπολέμηση της φτώχειας. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε με πολιτικές ε, βήμα προς βήμα. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε μια σφαιρική πολιτική στη βάση ενός σωστού προγραμματισμού αντιμετωπίζοντας τα μακροπρόθεσμα προβλήματα και τις μακροπρόθεσμες πολιτικές επιλογές. Τέταρτον, το ζήτημα του φίλου ε, είναι σημαντικό όσον αφορά τη χάραξη πολιτικών. Στη δική μου παρουσίαση μπορείτε να δείτε κάποια σχόλια σε σχέση με το θέμα αυτό από τη Φιλανδική Σκοπιά. Νομίζω ότι υπάρχει στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. Ο κίνδυνος της φτώχειας είναι μεγαλύτερος στις ηλικιωμένε γυναίκες που βασίζονται αποκλειστικά στη σύνταξή τους. Έχουμε και στη Φλανδία αυτή την ομάδα. Είναι ε, μικρή αλλά υπαρκτή και ορισμένες προσαρμογές μπορείτε να φανταστείτε τις ηλικιωμένες αυτές γυναίκες που έχουν μόνο αυτή τη βασική σύνταξη. εδώ ο κίνδυνος στόχιας είναι υψηλότερος. Ορισμένες προσαρμογές ε, ε, έχουν γίνει και ένα νέο σχέδιο νόμου ε, για, για το συνταξιοδοτικό θα ψηφιστεί το 2011, το Μάρτιο. Έχουμε προσπαθήσει λοιπόν να κάνουμε κάτι για να αντιστρέψουμε αυτή την τάση. Όσον αφορά τη φτώχεια των παιδιών, και εδώ βλέπουμε ότι η Φινλανδία σε σύγκριση με τι άλλε χώρε τα καταφέρνει αρκετά καλά. Ωστόσο, σε οικογένειε με χαμηλέ αποδοχέ υπάρχουν πολλά παιδιά και στη Φιλανδία. Οι χαμηλές αποδοχές απαντώνται πιο συχνά σε μονογονεϊκές οικογένειες όπου οι γυναίκες είναι συνήθως το γονεϊκό μέλος. Και αυτό ήταν και το συμπέρασμα σε μια πρόσφατη έρευνα για τη συντάξη των γυναικών που κάλυψε οκτώ χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αρχή παρουσίαση είχα κάνει μια σχετική μία, δεν θα να μπω εδώ σε λεπτομέρειες, αλλά σημειώνεται εδώ αυτό το, αυτή η κατάσταση στην οποία αναφέρθηκε άλλωστε και η προηγούμενη ομιλήτρια. Τα σχόλια μου λοιπόν βασίζονται στη φιλανδική εμπειρία, αλλά υποθέτω ότι έχουν, μπορούν να έχουν νόημα και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πριν, πριν κλείσω θα ήθελα να πω ότι ξεκινήσαμε με την προετοιμασία του δικού μας ε, προγράμματος μεταρρύθμισης για την, το 2020 Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, στοχεύοντας να δώσουμε μια σφαιρική φιλανδική απάντηση και ένα αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της απάντησης είναι ο στόχος καταπολέμησης της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. στοχεύουμε σε άνεργες οικογένειες, μακροπρόθεσμα άνεργους, με χαμηλές αποδοχές, συχνά μετανάστες και ειδικέ ομάδες επίσης. Αλλά δάδοντας κυρίως την έμφαση σε χάραξη ενεργών πολιτικών που δεν αφορούν τόσο πολύ τις υλικέ στερήσεις, γιατί στη Φιλανδία ε, το βλέπουμε αυτό που η διαφορά μεταξύ των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων, οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες μεταξύ των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων στη βάση αυτών των δικτών. Ανεργία και χαμηλές αποδοχές είναι η βασική διασύνδεση, το βασικό ζεύγος στο οποίο βασίζεται ο, το σχετικό νομοσχέδιο και ο προγραμματισμός στη Φιλανδία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κόχο από τη Φιλανδία. Πολύ σωστή ενημέρωση είχαμε από την τη Φιλανδία που αφορά τη έργο μας. Απλώς να σας πω εδώ κάτι. Ένα σχόλιο με αυτά που είπε ο κ. Κόχο ότι είναι ο μοναδικός άνδρας στις δύο πάνελ που είχαμε. Αυτό με κάνει να σχολιάσω ότι η πρώτη φορά που ανέλαβα κάτι πολιτικής φύσεως ήταν σε μια ε, επιχείρηση και εκεί πέρα βρέθηκα εγώ μοναδική γυναίκα ανάμεσα σε 50 άνδρες. Και, και γι' αυτό όλοι θεωρούσαν, πάρα πολλοί θεωρούσαν ότι εγώ πρέπει να ήμουν γραμματέας κάποιου από αυτούς του 50, 50 άνδρες. Τέλος πάντων, αυτά σαν ένα σχόλιο ανεκδοτολογικά. Τώρα, στη συνέχεια, να χαιρετήσω την κυρία Μύρια Βασιλιάδου, που είναι Γενική Γραμματέας για το λόμπι, τον ε, Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών. Καλώς ήρθατε εδώ σε εμά και σας δίνουμε αμέσως το λόγο. Παρακαλώ. Thank you very much. I hope you can... Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να με ανεχτείτε γιατί ήταν μακρύ το απόγευμα και είναι πάντα δύσκολο τέτοια ώρα. Ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση και ευχαριστώ όλα τα μέλη του πάνελ. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και καμιά φορά είναι δύσκολο να μην επαναλαμβάνονται θέματα. Απ' την άλλη βέβαια η εμπειρία μου σαν μέλος λόμπι είναι ότι είναι καλό να επαναλαμβάνεις πράγματα πολλές φορές. Κάτι που θα πρέπει να θυμηθούμε καταρχάς είναι ότι η φτώχεια, η βία και το να είναι κανείς άστεγος είναι αλληλένδετα και μπορεί να τα θεωρούμε αυτά σαν δεδομένα, η αλήθεια είναι ότι αυτέ οι σχέσει πρόσφατα έγιναν αποδεκτέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν μπει στο πρόγραμμα. Η σημερινή ακρόαση για μένα είναι πολύ τιμή, κυρίω για αυτόν τον λόγο. Και αν δεν καταλάβουμε αυτά τα θέματα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε την διάσταση του φύλου στην φτώχεια και πώ θα αντιμετωπίσουν οι γυναίκε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Κάθε φορά που αναφέρομαι στη φτώχεια, θα αναφέρομαι και στον κοινωνικό αποκλεισμό διότι όπως ακούσαμε και από άλλους ε, μιλητές δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων αλλά και προσβάσεως σε υπηρεσίες πολιτικής λήψεως αποφάσεων, να έχει κάνει μια φωνή, να έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε όλες τις πτυχές της ζωής. Άρα αφορά τις γυναίκες στο κάτω-κάτω της γραφής. Αυτό που προσπαθήσω να κάνω είναι να πω μερικά πράγματα για τη δουλειά που κάνουμε και να συναγάγω κάποια συμπεράσματα ποια είναι η σχέση μεταξύ γυναικών και φτώχεια στην Ευρώπη, ποια είναι τα βασικά ζητήματα και να καταλήξω ελπίζω σε κάποιες συστάσεις. Να υπενθυμίσω ότι είμαστε η μεγαλύτερη γενική οργάνωση. Έχουμε περίπου 2.500 μέλη, οργάνωση γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη και τρει υποψήφιε χώρε. Εξαιρείται η Ισλανδία για την ώρα. Τώρα, η δουλειά που κάνουμε για τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ε, φτώχεια ήταν αναπόσπαστο τμήμα η φτώχεια τη γυναίκα τη δουλειά που κάναμε όσον αφορά τι κοινωνικέ πολιτικέ και την απασχόληση. Υπήρξαμε ενεργά μέλη του συνασπισμού κοινωνικών μη κυβερνητικών οργανώσεων για το ευρωπαϊκό έτο 2010 για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη παινία. Το 2010 κάναμε μια δήλωση όσον τι γυναίκε και τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στα πλαίσια του έτου αυτού. Περαιτέρω, λόγω τη χρηματοστική κρίσης και λόγω του του ευρωπαϊκού έτου αυτού, η AWL και η Oxfam το Φεβράριο του 2010 εξέδωσαν μια κοινή έκθεση πολιτικής για τις συνέπειες που έχει η ύφεση στις γυναίκες και για τη φτώχεια. Και από τίτλο έχει «Η κρυμμένη κρίση». Θα αναφερθώ στο κρυμμένο αυτό στοιχείο. Αργότερα σε δύο εβδομάδες θα έχουμε νέα στο σελίδα και όλα αυτά θα είναι πολύ εύκολα να τα βρείτε. Τώρα, όσον αφορά την έκθεση που συντάξαμε μαζί με την Oxfam, δεν είναι κάτι που απλώς λέμε, είναι κάτι που τερευνήσαμε εκτενώς. Η φτώχεια έχει θηλυκό πρόσωπο. Και ο συνεχής περιθυροποίηση των γυναικών είναι συνεχές πρόβλημα που απορρέει από τις ανισότητες. Και η βάση της παρουσιάσεώς μου είναι αυτή, δηλαδή ότι είναι κάτι που άμεσα συνδέεται με τις ανισότητες. Όταν πλειοψηφία των γυναικών Ρώμα στη Βουλγαρία γεννούν σε σπίτια χωρίς τρεχούμενο νερό ενώ κάποιες προνομιούχο στη Ρουμανία υπάρχουν. Εμεί ένας μου στο γραφείο γέννησε με ευτήριο, αλλά ήταν διαφορετικό με ευτήριο από τις ε, ευτήριο πάνω στις γυναίες και στη Ρουμανία. Υπάρχει διαχωρισμός. Λοιπόν, υπάρχουν σοβαρέ ανισότητες, όπου οι γυναίκες είναι τέσσερις φορές πιθανότερο να εργαστούν σε μερική απασχόληση για να ε, ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του στα νοικοκυριά. Υπάρχουν και άλλα πορίσματα βεβαίω που περιέχονται στην της και οι γυναίκες χάνουν τη δουλειά τους και τα εισοδήματά τους. Όλοι κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Αλλά ποιο χάνει τι. Αυτό εξαρτάται από την ε, δομή της οικονομίας και το βαθμό στον οποίο οι πολιτικές ε, ε, εθελοτυφλούν όσον αφορά το φύλλο, τη διάσταση του φύλλου. Και ποιε είναι οι συνέπειε όσον αφορά τι γυναίκε αν γέννη και ποιοι γίνεται με τα μέλη των ευαλώτων ομάδων που αντιμετωπίζουν πολλαπλά μειονεκτήματα. Εκεί συμπεριλαμβάνονται οι ηλικιωμένε, οι νέε, οι εθνικέ μειονότητε, οι μετανάστε, αυτέ που δεν έχουν δεξιότητε, αυτέ που έχουν συμβάσει μικρά δια... διαρκεία. Και έχουμε ένα μακροσκελή κατάλογο προβληματικών ομάδων. Και είδαμε ότι οι μειώσει στι δημόσιε δαπάνε πάντα θα έχουν σημαντικέ και δυσανάλογε συνέπειε για, την... Ε, για των γυναικών. Οι γυναίκε είναι στον τομέα, κυρίω στο δημόσιο τομέα, στην πλειοψηφία του. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 80% οικοδόμων είναι άντρε 78% στις κοινωνικές υπηρεσίες και στην πρόνοια είναι γυναίκες. 60% των δασκάλων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι γυναίκες και εκεί έχουν γίνει μεγαλύτερε περικοπές. Ας ρίξουμε μια ματιά λοιπόν σε αυτό το χάρτη. Όπως είπα, η φτώχεια δεν αφορά μόνο τα χρήματα, αλλά αφορά και το να είναι κανεί άστεγος, να μην έχει δυνατότητε, έλλειψη πρόσβαση ε, στην υγιή διατροφή κλπ. κλπ. Όμως οι στρατηγικέ της Ευρωπαϊκή Πολιτική δεν συμπεριλαμβάνουν την, σαν στόχο την ισότητα των φύλων και η συμπερίληψη της, του διάσταση του φύλου στις πολιτικές παραμένει κάτι πολύ ισχνό. Λοιπόν, μετανάστευση, ε, καταπολέμηση του εμπορίου ε, ε, ανθρώπων είναι κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το είπαν και από το WAVE και το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα σε αυτό το θέμα. Ο κοινωνικό αποκλεισμό και η φτώχεια οδηγεί σε κακή στέγαση στι γυναίκε. Καμιά φορά να ζουν στου δρόμου οι γυναίκε και στη βία καμιά φορά. Περαιτέρω βία και άλλη βία. Οδηγεί στην πορνεία, οδηγεί στο εμπόριο του σεξ. Όλα αυτά τα θέματα ε, τα ανέφεραν οι προελίσσαντες. Δεν θα επισταθώ σε λεπτομέρειες, αλλά η διαφορά των εισοδημάτων των φύλων, όπως αναφέρθηκε, αυτό το κενό είναι σημαντικό πρόβλημα. Εκεί ε, βλέπουμε πώς οι γυναίκες μπορούν να καταλήξουν φτωχές ή να κινδυνεύουν να ζουν στη φτώχεια. Να υπενθυμίσω σε όλες ότι η ισότιμη αμοιβή αναφέρθηκε πρώτα φορά το 57 και είμαστε αυτή την αίθουσα σήμερα και μιλάμε για τη διαφορά της αμοιβή των φύλων. 50 χρόνια αργότερα μιλάμε ε, για αυτό το θέμα. Και είναι παραπλανητικό αν δούμε απλώ το φορολογικό έτος και τη χρήση αυτή και λέμε η Ιταλία τα πάει καλά, κοιτάξτε τι γίνεται με την Τσεχία. Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι της εικόνας, αλλά δεν είναι η εικόνα στο σύνολό της. Παραδείγματο χάρη, η διαφορά των αμοιβών αφορά τι γυναίκε όλου του τομεί τη αγορά εργασία, αλλά κυρίω αυτέ που δεν έχουν δεξιότητε, όπω είναι η παροχή υπηρεσιών, φροντίδα, που έχουν ε, συμβάσεις μικρής διαρκείας ορισμένου χρόνου. Λοιπόν, οι γυναίκες που φροντίζουν ηλικιωμένου βγάζουν λιγότερο από έναν άντρα που είναι οικοδόμος ή εργάζεται στην ε, μεταποιητική βιομηχανία. Και αυτό αφορά το θέμα της φροντίδας. Ποιος φροντίζει, ποιος παρέχει τη φροντίδα. Αυτό είναι ένα κομμάτι της ε, εκστατείας μας πριν από τρία χρόνια. Η προσδοκία αφορά τη φροντίδα και πώς το συνδέουμε αυτό με τη διαφορά, της τη διαφορά των φύλων. Διότι πρέπει να δούμε και ποια είναι η φύση της φροντίδας. Κοιτάξτε τις εικόνες που σας δείχνω. Ελπίζω να φαίνονται. Βλέπετε εδώ στην οθόνη τις εικόνες. Είναι έρευνα του Google. ηλικιωμένες, φροντίδα ηλικιωμένων και παιδιών. Τα στερεότυπα υπάρχουν παντού. Ε, ποιότητα και ευθυνή μέρημνα. Είναι κάτι που δεν ε, καλύπτεται ιδιαίτερα. Σε κάποιε χώρε, όπω οι σκανδιναβικέ χώρε, τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Η τσεχική δημοκρατία έχει 80% των γυναικών που εργάζονται με μερική απασχόληση, ούτω ώστε να ασχοληθούν με τι ευθύνε του όσον αφορά τη φροντίδα. Αυτό δεν φαίνεται εκεί. Αλλά δεν σε εκπλήσει ότι στη τσεχική δημοκρατία έχουμε τόσο υψηλό ποσοστό διαφορά αμοιβών ανάλογα με το φύλλο. Μετά η Ένωση δεν ανταποκρίθηκε στους στόχους της Βαρκελόνης για τη φροντίδα των παιδιών. Τώρα να αλλάξω χάρτη. Όπως και να δούμε το χάρτη και την εικόνα, όποιο σχήμα και αν δώσουμε σε αυτά τα στοιχεία τα αριθμητικά, πάντα το ίδιο είναι το ζουμί. Οι γυναίκες είναι πιθανότερο να πληγούν από τη φτώχεια από ότι άντρες. Ακούσαμε τώρα τις διάφορες ομάδες που αναφέρθηκαν. Πώ πλήττονται σε διαφορετικό βαθμό ανάλογα με την ομάδα από τη φτώχεια. Τι διακυβεύεται εδώ. Και θα επανέλθω σε αυτό που είπα στην αρχή τώρα. Η ανισότητα. Περί αυτού πρόκειται. Και είναι ισότητα με βάση το φύλλο. Και αυτές είναι οι πιο ευρέω διαδεδομένες μορφές ανισότητας που βλέπουμε στην αγορά εργασία με τη διαφορά των αμοιβών. Το βλέπουμε πιο γενικά στον πολιτισμό και στην οτροπία. Με με όσον αφορά τις εταιρείε που δεν ανεβαίνουν στα νότερα αξιώματα οι γυναίκε. κολλάνε στο πάτωμα αν θέλετε. Το βλέπουμε στο νόμο για διζυγία, φορολογία, κοινωνική προστασία, συντάξει. Ε, η Αν Σοφή είπε καλύτερα από μένα. Λοιπόν και το χειρότερο είναι ότι αυτές οι ανισότητες με βάση το φύλλο επηρεάζουν και υπάρχει αλληλεπίδραση και με άλλου παράγοντε. Και πάμε στο κρυμμένο πρόσωπο τη φτώχεια. Μιλήσαμε για το πώ είναι αόρατη η βία κατά των γυναικών όσον αφορά τη φτώχεια, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που είναι αόρατο, οι νομικές ανισότητες. Ε, και εδώ κρύβεται η φτώχεια των γυναικών. Τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να υπολογίζουν τη φτώχεια επί τη βάση σορευμένου συνολικού εισοδήματο των οικοκυριών, Υποθέτοντα ότι και και γυναίκα βγάζουν τα ίδια και κατανέμουν εξίσου του πόρου. Όλα ωραία και καλά ε, ε, ε, οι γυναίκε εξακολουθούν να δουλεύουν στο σπίτι και να μην αμείβονται και να φροντίζουν και να μην αμείβονται. Και αυτό δεν υπολογίζεται στου στι συντάξει. Και αν πεθάνει ο σύντροφο ή αν χωρίσουν από τον σύντροφο, κινδυνεύουν να μπουν στη φτώχεια οι γυναίκε. Χρειαζόμαστε ατομικά δικαιώματα και πρέπει να υπολογίζουμε τα ατομικά εισοδήματα. Όπω βλέπετε στα δεξιά του γραφήματο, τα αποτελέσματα θα ήταν εκπληκτικά να ξεκινούσαμε του υπολογισμού. Θα πρέπει. Στο 36% είναι ο πραγματικό κίνδυνο για τη γυναίκε. Για τους άντρες είναι κάτω, είναι 11%. Δεν θα πω τίποτα για τις συντάξει, νομίζω ότι με κάλυψε η Αν Σοφή και θα ήθελα να πω ότι εμείς θέλουμε να εργαστούμε σε αυτό το τομέα, συνεργαζόμαστε με την πλατφόρμα, την H Platform και βλέπουμε τι γίνεται και με την πράσινη βίβλο για τις συντάξει που θα ξέρετε. Ας πω και σε κάτι άλλο που είναι αόρατο τώρα. Οι γυναίκες και το να είναι άστεγες η έλλειψη στέγαση. Θα ξεκινήσω τώρα από τις εικόνες, Μ' αρέσουν οι εικόνε. Κοιτάξτε την εικόνα. Εδώ βλέπουμε πώ φαίνεται ποιο είναι ένα, ένας άστεγος, ένας στον πάγκο. Αλλά το μήνυμα ποιο είναι, ότι οι άστεγοι είναι άντρε, πρώτον, και ότι είναι μειοψηφία οι άστεγοι στον δρόμο, διότι οι περισσότερε όμω ζουν σε κρυμμένα, ε, ε, κρυπτό είναι άστεγες. Μπορούν να μείνουν με φίλους, με οικογένειες, με γνωστούς, και κινδυνεύουν το τρόπος περισσότερο όσον αφορά την εκμετάλλευση με τη, έναντι της βίας και χάνουν και δικαιώματα όσον αφορά την υποστήριξή τους. Αν βρούνε βραχυπρόθεσμη στέγαση, οι κοινωνικές υπηρεσίες τους μη θεωρούν ως άστεγες και τους αρνούνται υποστήριξη. Κρύβονται με την νομική έννοια του όρου. Κρύβονται όσον αφορά τη βία, κρύβονται όσον αφορά το πρόβλημα της στέγασης, όταν μένουν άστεγες. Και κάτι που θα πρέπει να εξετάζουμε και να προσέξουμε και έχουμε σχετικά κάποιο δημοσίευμα είναι ο διαλειτουργικός χαρακτήρας, διατομικός χαρακτήρας της ανισότητας των φύλων όπου το φύλλο ε, συντονίζεται με άλλες μορφές διάκρισης και ανισοτήτων. Αναφέραμε Κροθυγό ένα παράδειγμα, μετανάστριες. Πολύ συχνά υποχρεούνται να ζουν στην ε, γκρίζα οικονομία, δεν έχουν συμβάσεις, εξαρτώνται από τους εργοδότες τους πιθανότατα. Αυτές οι γυναίκες εργάζονται σε θέσεις προσωρινές, άρα αποκλείονται από τις κοινωνικές εισφορές, ε, άδεια αγωνική, ε, μητρική άδεια κλπ. Και κάποιες και δεν έχουν και νομικό καθεστώς να είναι στην Ένωση, διότι έχουν εξαρτώμενο νομικό καθεστώς. Αυτό προαναφέρθηκε και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να εξεταστεί. Και ένας άλλος τρόπος που βλέπουμε αυτή την αλληλεπίδραση των διαφορών παραγόντων. Αν δούμε τι γίνεται, γυναίκες με τις Ρώμα, το φίλο με τους Ρώμα, πώς συνδέεται. Είναι τόσο περιοθυροποιημένες, το ακούμε γιατί είναι της μόδας τελευταίες δύο εβδομάδες. Αλλά αυτή δεν είναι κατάσταση πρόβλημα δύο εβδομάδων. Είναι δύσκολο να βρει κανείς στατιστικά στοιχεία που να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα των γυναικών Ρώμα. Αν επαρκεί στέγαση, ε, μένουν έγκυες όταν είναι έφηβες, υπάρχει μεγάλη ανεργία, δεν υπάρχει επαρκής ε, περίθαλψη κλπ. Όλα αυτά αφορά η φτώχεια. Έχουμε λοιπόν κάποια στατιστικά στοιχεία και σίγουρα δεν αρκούν. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ξανά ότι οι γυναίκες που είναι 52% του πληθυσμού της Ευρώπης υπόκειται σε πολλαπλά επίπεδα ε, διάκρισης που έχουν αλληλεπίδραση μεταξύ τους αυτές οι πτυχές της διάκρισης. Τι βλέπουμε λοιπόν. Υπάρχουν άλλοι που είναι καλύτεροι από μένα να αναφερθούν στο πρόγραμμα του 2020 και έχουμε το προηγούμενο μέλος του πάνελ που αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Όμως, είναι το πρώτο ευρωπαϊκό έγγραφο, ελπίζω να μην σφάλω, που έχει ένα ποιοτικό στόχο, την εξάλληψη της παινίας. Το πρώτο έγγραφο. Χρειαζόμαστε τη διάσταση του φύλου στο στόχο αυτό κατά πολέμηση Είναι απόλυτα αναγκαίο. Έχουμε 75% στόχο απασχόληση για τι γυναίκε. Αυτό δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί αν δεν ληφθεί υπόψη γενικότερα το όλο φάσμα των γυναικών. Τι γίνεται με τη διαφορά των αμοιβών, part-time, ευέλικτη επασχόληση, άλλε στοιχείε τη ζωή τη γυναίκα, αν δεν ληφθούν υπόψη, το 75% λέει ελάχιστα για μένα, αν λέει και κάτι. Δεν έχει νόημα δηλαδή. Ε, βέβαια, έχουμε και την μέθοδο ανοιχτού συντονισμού και εδώ τα κράτη-μέλη πράγματι μπορούν να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές για κοινωνικά ζητήματα. Έχουμε τα διαθροτικά ταμεία, τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας με τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Υπάρχει μια ισχυρή νομική βάση, πιστεύω, για την καταπολέμηση της στόχιας. Ε, είναι και ισχυρό νομικό και ηθικό, το τονίζω εργαλείο στα χέρια εκείνων που παίρνουν τι αποφάσει στι πολιτικέ. Και έχουμε και το Ευρωπαϊκό Έτο και θέλω να τονίσω ότι έχουμε όλα αυτά τα εργαλεία και αυτό που χρειαζόμαστε είναι να θυμόμαστε πάντα ότι χρειάζεται ατομικά δικαιώματα όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και τι συντάξει. Οι γυναίκε εξαρτώνται από αυτά τα συστήματα. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να το θέσουμε. Και το κράτο δεν θα πρέπει να αντικαθιστά τον άντρα και τον σύντροφο σε αυτά τα συστήματα. Στην τελευταία μου διαφάνεια, και είναι η τελευταία διαφάνεια αυτή, θα πω ότι σήμερα τρόπο βγήκε ένα μήνυμα ότι η φτώχεια έχει θηλυκό πρόσωπο και ότι η συνεχής οικονομική περιφερειοποίηση των γυναικών είναι ένα επίμονο πρόβλημα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Αναφέρθηκα στις ρίζες του κακού. Μπορούμε να το αναφέρουμε επανειλημμένα, αλλά τα εργαλεία που έχουμε, τα είδαμε στην προηγούμενη διαφάνεια. Τι μου λένε αυτά τα εργαλεία, ότι υπάρχει ένα πράγμα που δεν έχουμε. Έχουμε τα εργαλεία, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, Κάποιοι λένε έχουμε αρκετούς στόχους, κάποιοι λένε δεν έχουμε αρκετούς. Δεν έχουμε πολιτική δέσμευση. Αυτό είναι σαφές από το 1957 όταν αναφέρθηκε η ίση αμοιβή. Αυτό είναι ξεκάθαρο για μένα. Έχουμε μία σύνοψη με κάποιες συστάσεις και σας διαθέτουμε πολλά έγγραφα. Δεν θα έχω, ε, δεν θα ετοιμάσω κατάλογο μακροσκελή συστάσεων, υπάρχουν. Κλείνοντα, να πω μερικά λόγια με μία από τι συστάσει όσον αφορά το πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάποιο ευρωβουλευτή που έφυγε το ανέφερε αυτό. Κάποια ευρωβουλευτή. Κάποιοι θα έλεγαν ότι οι περισσότεροι φτωχοί στον κόσμο είναι γυναίκε και αυτό ίσω δεν μπορεί να υποστηριχθεί. Πώ το ξέρει κανεί, πού είναι τα στατιστικά στοιχεία. Η μειονεκτική θέση των γυναικών όμω είναι κάτι αδιαφυσβήτητο. Υποφέρουν από τη φτώχεια με πολλαπλό τρόπο. Είναι σε δυσμενή θέση εναντί των ανδρών και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Εργάζονται πιο πολύ και στην παραγωγική δραστηριότητα και την αναπαραγωγική δραστηριότητα και βγάζουν λιγότερα χρήματα. Αυτό είναι γεγονό. Η δυνατότητα να μείνουν εκτό φτώχεια μπλοκάρεται από θέματα αγορά-εργασία, πολιτιστικά, ε, οικονομικά κλπ. Και κρύβονται διάφορε συνθήκε. Αυτέ επιδεινώνται συνθήκε από το περιβάλλον τη νεοφιλελεύθερη πολιτική και την ανακατανομή των πόρων. Για αυτού του λόγου η φτώχεια ίσω να είναι πλέον χρόνια μεταξύ γυναικών και πιο περαστική μεταξύ ανδρών. Και αυτό είναι κάτι άλλο που πρέπει να θυμόμαστε. Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να βγει σαν μήνυμα εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λόμπι για τις γυναίκε, είναι ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, η υλοποίησή του, και η ενίσχυση των γυναικών είναι βασικό συστατικό τη ευρύτερη διαπάλης κατά τη φτώχεια. Αυτό είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Πολιτική δέσμευση, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε πιστεύω. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βασιλιάδου. Σας ευχαριστούμε κύριε Βασιλιάδου λοιπόν για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση με όλες τις πληροφορίες που λάβαμε. Όλα είναι ξεκάθαρα και τώρα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε σχολιασμό από τις συναδέρφους. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπάρμπαρα Ματέρα, η οποία είναι σκιώδης εισηγήτρια και ανήκει Στου χριστιανοδημοκράτε, στην πολιτική ομάδα του Κοινοβουλίου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, έτσι έλεγε στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών που τελείωσε στη Νέα Υόρκη και διεξήχθη στη Νέα Υόρκη και επιβεβαίωσε τους στόχους της χιλιετίας. Ο πρώτος και πιο σημαντικός στόχος είναι να εξαλειφθεί η ακραία φτώχεια, η πείνα αλλά και να εγγυηθούμε την παιδεία, την ισότητα των φίλων, την... να καταπολεμηθεί η θνησιμότητα των παιδιών, να βελτιωθεί η υγεία των παιδιών, να καταπολεμηθούν διάφορε σοβαρέ ασθένειε και να υπάρχει περιβαλλοντική βιωσιμότητα και να προωθηθεί η ανάπτυξη. Οκτώ θεμελιώδη σημεία που υπόγραψαν περίπου 200 χώρε και πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2015. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή είναι μια αναφορά ε, στην ε, διάσκεψη του ΟΗΕ Σκεφτείτε ότι στην η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό ποσοστό των χωρών που υπέγραψαν αυτά τα σημεία που προανέφερα και εμείς εδώ σήμερα ε, μιλάμε για γενικούς στόχους, παγκόσμιους στόχους και λοιπόν μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι γραμμές που θα μας προσανατολίσουν και που θα μας οδηγήσουν να συντονιστούμε τη άσκεψη της Νέας Υόρκης. Μια μάχη με τη φτώχεια που είναι αδιαφυσβήτητα μια προτεραιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε αυτή τη μάχη μεταξύ των στόχων της στρατηγικής για το 2020 όπως επανειλημμένα ακούσαμε. Ε, ο ΙΕ σε παγκόσμιο επίπεδο άφησε πέντε χρόνια μπροστά μας για να μειωθεί σημαντικά αυτό το πρόβλημα. Εμείς εδώ σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να προτείνουμε τις στρατηγικές και τη διαδρομή που είναι καλύτερη. Η φτώχεια λοιπόν είναι ε, ε, αίτιο και δημιουργεί βία. Ε, κοινωνική απομόνωση, διάκριση και εξάρτηση έναντι των ανδρών. Ε, πιστεύω ότι είναι η δική μας αρμοδιότητα και καθήκον να προσθέσουμε να δώσουμε ζωή σε πολιτικές που προστατεύουν τις γυναίκες και πάνω απ' όλα όσον αφορά το κοινωνικό τους, την κοινωνική τους θέση. Μετανάστριες ε, που είναι πιο ευάλωτες, κυρίως γιατί είναι μόνες τους και με παιδιά, χωρίς δουλειά ή με πρόβλημα για να μπορέσουν να βρουν κάποια δουλειά οι γυναίκες που είναι υποχρεωμένες να, επι... να διαλέξουν part-time μερική απασχόληση είναι χωρίς στέγαση, χωρίς κοινωνική αρρωγή, με ελάχιστη βοήθεια όσον αφορά την ε, υγειονομική προστασία. Ε, ε, πληρώνουν την οικονομική κρίση και στις χώρες μας. Δεν μιλάμε για γυναίκες υπό ανά των χωρών, μιλάμε για γυναίκες τώρα που είναι ε, γυναίκες κόρες των, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Ευρωπαί, Ευρωπαίες γυναίκες μιλάμε σήμερα και αναφερόμαστε σε γυναίκες που ασχολούνται σε δραστηριότητες στην Ήπεθρο που δεν αναγνωρίζονται και που είναι αντικείμενα εκμετάλλευσης. Είναι και γυναίκες που δεν μπορούν να εγγυηθούν το μέλλον τους, διότι δεν καταφέρουν να φτάσουν ούτε στο αύριο, να δουν θα γίνει αύριο. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια φωνή σε όλες αυτές τις γυναίκες που θα αποφασίσουν να μιλήσουν και θα πρέπει να συμμετάσχει η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να εμπλακούν οι διάφορες οργανώσεις, οι ενώσεις και κυρίως τα πανεπιστήμια, πάνω από όλα τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Πρέπει λοιπόν να εγγυηθούμε στο να ότι θα εισακωστούν αυτές οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν δυσκολίε. Να υπάρχει ένα πράσινο νούμερο τηλεφωνικό που θα εγγυάται βοήθεια όσον αφορά την υγεία, τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματά τους θα πρέπει αυτά τα κέντρα τηλεφωνικά να είναι άμεση επαφή με τα Υπουργεία των 27 κρατών μελών, να μπορούν να μιλάνε όλες τις γλώσσες που είναι γνωστές. Διαφορετικά η δημιουργία αυτού του πράσινου αριθμού θα είναι εισμάτιν. Θα πρέπει να προωθηθεί μια σειρά μελετών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα παρακολουθούν και τις ανάγκες που έχουν οι γυναίκες οι ηλικιωμένες όσον αφορά την κοινωνική αρρωγή και υγειονομική αρρωγή που θα παρέχεται δωρεάν θα πρέπει να ζητήσουμε τα κράτη-μέλη να παρέχουν και κατοίκον πρόνοια και για του φτωχού και για τα άτομα που ε, δεν μπορούν να μετακινηθούν. Με αναπηρία θα πρέπει να δημιουργηθεί δυνατότητα εργασία, να αξιολογηθεί, να αξιοποιηθεί η δουλειά των γυναικών, δίνοντα κυρίω να δώσουμε κίνητρα στι γυναίκε που είναι νέε και στι γυναίκε που είναι πιο ηλικιωμένε να καλυφθούν. Φτάνω σύντομα στα συμπεράσματα. Πρέπει να αγγιθούμε την δωρεάν νομική αρρωγή σε αυτές τις γυναίκες όπου τις βιάζουν οι, γυναί... Ε, οι σύντροφοί τους και τι γίνεται με την ε, ε, ανατροφή των παιδιών. Θα πρέπει να δοθεί νομική βοήθεια δωρεάν σε περίπτωση άδικης απόλυσης, σε περίπτωση φυσικής ή ψυχολογικής βίας εκτός ή εντός των τείχων του σπιτιού. Για ακόμα μια φορά θα ήθελα να προσλαμβάνονται, να υπάρχει κινήτρο να προσλαμβάνονται γυναίκες που έχουν παιδί ακόμα και αν είναι μεγάλες ηλικία. Ε, θα πρέπει στην Ευρώπη να αναγνωρίζεται και να αξιοποιείται η λειτουργία του πολιτισμικού διαμεσολαβητή, κυρίως για τις μετανάστριες ε, γυναίκες. Θα έλεγα ότι όσον αφορά την αρχή της επικουρικότητας, δεν μπορούμε να μην προσέξουμε και να υποστηρίξουμε τις πολιτικές εκείνες να δοθεί νέα διάσταση πρόθεση, να τονιστεί η φτώχεια των γυναικών. Οι γυναίκες είναι η καρδιά της κοινωνίας, πέραν το ότι είναι και η καρδιά όλων των οικογενειών, σε όλες τις οικογένειες του κόσμου. Ευχαριστούμε την κυρία Ματέρα. Αμέσως μετά η κυρία Φιγκερέντο, η οποία είναι και αυτή η σκιώδης ισχυήτρια και ανήκει στην ομοσπονδιακή ομάδα την Ευρωπαϊκή Αριστερά, την ΚΟΥΗ. Την ΚΟΥΗ. Θα παρακαλώ, θα τη δώσουμε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Ε, numa hora muito avançada da nossa ε, discussão, e eu queria começar apenas por sublinhar três questões. Θα ήθελα να θέσω τρία ερωτήματα. Πρώτον, ε, το 2011 το, το 2010 είναι το ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της ε, φτώχειας, όπως ήδη υπόθηκε και προσπαθούμε μέσω αυτής της ε, δράσης να πετύχουμε μεγαλύτερη ορατότητα. Ε, ζητούμε την εξάλληση ελάχιστων αποδοχών για την καταπολέμηση της φτώχειας και για τον, την καλύτερη κοινωνική ένταξη. Εγώ είμαι η συγγήτρια αυτής της έκθεσης και η έκθεση αυτή θα συζητηθεί στις 18 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο. Η σχετική ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 20 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο. Θα ήθελα στο πλαίσιο αυτό να αναφερθώ σε διάφορα θέματα. Φυσικά θα επαναλάβω κάποια πράγματα τα οποία ήδη έχουν υποθεί, ωστόσο τα σημεία αυτά μου φαίνονται σημαντικά. Καταρχήν όσον αφορά την, το πολιτικό τομέα εν γέννη. Ο Φιλανδός Προσκακλημένος αναφέρθηκε σχετικά γιατί αυτό είναι ένα κεντρικό θέμα όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας. Το ζήτημα της πολιτικής δηλαδή. Εάν δεν προσδώσουμε αντίστοιχη σημασία στην σφαιρική πολιτική, θα εκπνεύσει το 2010 και θα υπάρξουν περισσότεροι φτωχοί ε, πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο ποτέ στο παρελθόν. Παρόλο που, όπως είπαμε, το 2010 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας. Και, όπως είπα, οι αριθμοί αυτοί θα είναι πρωτόγνωροι και πλήττουν κυρίως τις γυναίκες. Οι, τα στοιχεία που έχουμε προέρχονται από το 2008. Το 2008 είχε αρχίσει ήδη να διαφαίνεται αυτή η τάση. Αλλά συγκεκριμένα η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί στις διάφορες χώρες και είναι δυνατόν με το τέλος του χρόνου να φτάσουμε σε αριθμούς ρεκόρ και φανεί πρωτόγνωρα στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό των ανθρώπων που πλήττονται από το φαινόμενο της φτώχειας. Ποιοι είναι οι λόγοι γι' αυτό. Η παγκόσμια πολιτική καταρχήν, η ευρωπαϊκή πολιτική εφαρμόζει μια πολιτική η οποία δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη σε αυτή την κατάσταση. Αντίθετα, η φτώχεια όλο ένα επιδεινούται, βαίνει επιδεινούμενη έχουμε τα λεγόμενα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας και τα κριτήρια αυτά χρησιμοποιούνται από τις χώρες μέλη, την Κομισιόν και το Συμβούλιο για να προωθήσουν τελικά κοινωνικές περικοπές. Ε, πρωτίστως γίνονται οικονομίες περικόπτοντας ε, υπηρεσίες ε, κοινής ωφέλειας και με τον τρόπο αυτό βεβαίως διονγκώνεται το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Έχουμε αύξηση της φτώχειας και των διακρίσεων. Και γι' αυτό θα βιώσουμε την δυνότερη κατάσταση των τελευταίων δεκαετιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το θεσπίστηκε ακριβώς αυτό το έτος 2010 ε, την καταπολέμηση της φτώχειας. Όταν λοιπόν λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και μια κοινωνική διάσταση, ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να αλλάξει αντίστοιχα και η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική. Και τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο τη προσοχή μα ω προτεραιότητε. Αλλιώ παραμένουν κενά λόγια τα οποία δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Αυτή είναι η λεγόμενη αφιλεύθερη πολιτική του Συμφώνου Σταθερότητας, η απελευθέρωση της ανεργίας κλπ. Η με περισσότερη απελευθέρωση, συγγνώμη, αύξηση της ανεργίας κλπ. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, τα ξέρουμε όλοι. Και στο πλαίσιο αυτό, τόσο η Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο, καθώς και οι χώρες μέλη, έχουν τώρα τη δυνατότητα να λάβουν κάποιες αποφάσεις. Κατά πόσο δηλαδή θα απεσταδρομήσουν ή θα είναι διατεθειμένες οι χώρες να ανταπακριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις εφόσον επιδεινωθεί η κατάσταση αυτή και αυξηθούν οι κοινωνικές εντάσεις. Κάτι που είναι πολύ πιθανό. Και στην περίπτωση αυτή βεβαίως θα μειωθεί και η εξοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις ε, προτάσεις που έχει κάνει για την ε, οικονομική και κοινωνική συνοχή. Αυτό είναι το βασικό θέμα της έκθεσης και πέρα από αυτό θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονός είναι σημαντικό να έχουμε θέσεις εργασίες που συνοδεύει, κατοχυρώνονται μέσω κάποιων δικαιωμάτων, γιατί υπάρχουν όλο και περισσότερες φτωχές γυναίκες κυρίως, που δεν έχουν ε, τέτοια εισοδήματα που θα μπορούσαν να τις απελευθερώσουν από αυτή την κατάσταση φτώχειας. Επισφαλείς ε, συνθήκες εργασίας, επαραδείγματι. Και αυτό είναι ένα κεντρικό θέμα. Όπως είπα λοιπόν, θα πρέπει οι θέσεις εργασίας να κατοχυρώνονται με σχετικά δικαιώματα και να αμείβονται αντίστοιχα. Πέρα από αυτό, ε, το ζητούμενο είναι ποιοτικέ υπηρεσίε, κοινή ωφέλεια, κοινωνική πρόνοια κλπ. Και επίση κατοχήρωση ενό ε, ελάχιστου ορίου αποδοχών για εκείνους που δεν έχουν άλλες ε, δυνατότητε, άλλου πόρους. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι τμήμα της πολιτικής μας. Η εξασφάλιση ελάχιστων αποδοχών που να ανταποκρίνονται στο κατόφλιο της φτώχειας. Η πρόεδρος διακόπτη. Ε, σας ευχαριστούμε. Τώρα θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Επιτροπής, η κυρία Μαριάν Παρασκευά. Έχει το λόγο, παρακαλώ. I will uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Ε, θα ήθελα να τονίσω κάποια σημεία που αναφέρθηκαν Πρώτα απ' όλα, όπως προανέφερα, ατομικά κοινωνικά δικαιώματα είναι ένα θέμα το οποίο το επεξεργάστηκε πριν από 15 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά το εγκαταλείφθη, οπότε θεωρώ ότι τώρα είναι η σωστή στιγμή να επανέλθουμε στο θέμα αυτό και παρομοίως θα ήθελα να αναφερθώ σε μια διάσκεψη που έλαβε χώρα περασμένη, την περασμένη Παρασκευή και διοργάνωση το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καταπολέμησης Φτώχειας για το ελάχιστο εισόδημα, όπου απευθύνθη έκκληση για εξατομικευμένο ελάχιστο εισόδημα που θα εκάλυπτε τον κύκλο ζωής, δηλαδή θα κάλυπτε και παιδιά, και παιδιά ε, άτομα ηλικίας εργάσιμης, είτε είχαν δυνατότητα να εργαστούν είτε όχι, και ηλικιωμένους. Αυτή ήταν μια έκκληση η οποία θα διαβιβαστεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Το θέμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αυτά είναι αλληλένδετα ζητήματα και γι' αυτό ο στόχος δεν είναι στόχος που αφορά μόνο τη φτώχεια, είναι ένας στόχος που αφορά και την πρόληψη, η καταπολέμηση της στόχιας του κοινωνικού αποκλεισμού επίσης και η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα θα, θα εστιαστεί όχι μόνο επί της φτώχειας αλλά και του κοινωνικού αποκλεισμού επίσης. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Αυτά τα δύο ζητήματα συνδέονται στενά με την μη διάκριση. Και με τις δυνατότητες που παρέχει η νέα συνθήκη τώρα, υπάρχει δυνατότητα να διερευνηθούν και αυτοί οι τομείς. Βέβαια, το ζήτημα της βίας και το εμπορίο λευκής σαρκός είναι κάτι που αναφέρθηκε εκ νέου. Εγώ θα ήθελα να συμπεριληφθούν στον τομέα της κοινωνικής εντάξεως και της καταπολεμήσεως της παινίας, όμως μέχρι τώρα δεν κατέστη δυνατόν. Όσον αφορά τους στόχους της Βαρκελόνης για τη φροντίδα των παιδιών, δεν θέλουμε μόνο να έχουμε επαρκείς τόπους για τη μέρημνα των παιδιών, αλλά και ποιοτικά κέντρα και χρηματοδοτήσαμε και ένα πρόγραμμα στα πλαίσια της πτυχής κοινωνικής ένταξης του Progress για την ποιότητα του εργατικού δυναμικού που θα πρέπει να είναι διαθέσιμο. Και αυτό αφορούσε μόνο τη μέρημνα των παιδιών. Και στα πλαίσια της στρατηγικής για την ισότητα των φύλων, αυτό είναι κάτι που θα επεκταθεί για να καλύψει και την ποιότητα της φροντίδας που απαιτείται και για τους ηλικιωμένους. Τι άλλο. Α, τώρα με τη νέα πλατφόρμα κατά πολεμήσεως του κοινωνικού αποκλεισμού και της παινίας και τα θέματα των φίλων θα, των φίλων θα λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση πολιτικών και όπως προανέφερα θα εξετάσουμε και τις πιο ευάλωτες γυναίκες. Δηλαδή γυναίκες που είναι μέλη μονογονικής οικογένειας, μετανάστριες, μέλη μειονοτήτων, γυναίκες Ρώμα και ηλικιωμένε. Αυτά για την ώρα. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικότατα στα θέματα που ετέθησαν σήμερα. Ευχαριστώ. Καλώς. Σας ευχαριστούμε. Το λόγο εδώ στις συναδέλφες για κάποιες ερωτήσεις στο πάνελ. Εγώ προσωπικά μπορώ να κάνω επίσης κάποια. Ξέρετε, σήμερα φαίνεται να υπάρχει μια ανυπομονησία από τους από τις συναδέλφους και είναι φυσικό αυτό. Ε, το έχουν υπογραμμίσει πολλοί από τους καλεσμένους μας. Αυτά τα θέματα τα έχουμε συζητήσει τόσα και τόσα χρόνια και φανταστείτε ότι ακόμα τα συζητάμε. Ενώ συχνά διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να κάνουν κάποια αλλαγή τέλο πάντων σε αυτή την κατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι όταν μιλάμε για φτώχεια, αυτό που διαπιστώνουμε είναι, είναι ότι υπάρχει μια τάση όπου πλήττονται όλο και πιο πολλοί οι γυναίκες. Και αυτό είναι σοβαρό. Σήμερα, εδώ και στο δεύτερο πάνελ που είχαμε, για τις καλύτερες μεθόδες και τα μέτρα και καμιά φορά, ξέρετε, σκέφτομαι εγώ και λέω, γιατί δεν μπορούμε να διαπιστώνουμε ε, ποιες είναι οι καλύτερες μεθόδους, μέθοδοι που έχουν εφαρμοστεί στις χώρες μας. Γιατί δεν το συνειδητοποιούμε, για να μπορέσουμε ενδεχομένως να μεταφέρουμε τέλος πάντων αυτές τις μεθόδους σε εφαρμογή και στις άλλες χώρες, δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει πλέον αυτή η δυνατότητα και θα έπρεπε μάλλον να είμαστε θέση να το κάναμε. Επίσης στο πάνελ αναφέρθηκε το θέμα της ε, ατομικής αλέγμα εφαρμογή των διαφορετικών κοινωνικών συστημάτων. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι εγώ είμαι από τη Σουηδία, ξέρετε. Η μεγαλύτερη επιτυχία που είχαμε σε επίπεδα ισότητας ήταν στο τέλος της περκατίας του 50 είχαμε την ατομική ε, φορολόγηση το οποίο έδινε άλλες δυνατότητες πλέον για τις γυναίκες να δουλέψουν, να συμβάλλουν, να συμμετέχουν σαν φορολογούμενες αλλά να έχουν και το ατομικό δικαίωμα, την προσωπική τους ε, ασφάλιση, την ε, σύνταξη Γι' αυτό ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό που αναφέρατε κι εσείς εδώ για την εξατομίκευση. Επίσης, να πω ότι είπαμε πολλά για το δικαίωμα στην απασχόληση. Εννοείται, εννοείται ότι οι γυναίκες θα έχουν αυτό το δικαίωμα. Αλλά, συγχρόνως, να δούμε, δεν θα μείνει δικαίωμα στα χαρτιά, αλλά να εξασφαλίσουμε ε, προϋποθέσεις να εφαρμοστεί να υπάρχει δηλαδή μια σωστή υποδομή, φροντίδα για τα παιδιά, ε, φροντίδα για τους ηλικιωμένους και επίσης να πω ότι και τη δουλειά που κάνουν πολλές γυναίκες και στις οποίες δεν αμείβονται, να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες μέθοδοι που έχουμε ούτω ώστε η γυναίκα να μπορεί να κάνει μια τέτοια απλήρωτη θα λέγαμε εργασία με τον καλύτερο τρόπο. Είναι σαφές λοιπόν ότι πρέπει να περάσουμε σε συγκεκριμένα μέτρα και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε και την έκθεση Βιγκερέντο όπου έχουν γίνονται κάποιες ε, προτάσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν για να προχωρήσουμε για να μειώσουμε τη φτώχεια. Φτώχεια δεν, η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομία αλλά έχει και τις συνέπειες ότι οι γυναίκες δεν μπορούν πλήρως να ενταχθούν στην κοινωνική ζωή, ε, υπόκεινται σε καταχρήσεις, σε άνηση μεταχείριση. Υπάρχει το θέμα της εμπορίας, το λευκής σαρκός και τα λοιπά που τα έχουμε πει. Ε, θα πρέπει δηλαδή και με, τον, και με την αρμόδια η συγγετρία να δούμε πώς μπορέσουμε να προχωρήσουμε για να δούμε, να περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Δεν ξέρω, κάποιος άλλος. Παρακαλώ, παρακαλώ, έχετε το λόγο να κάνετε σχόλια. Ε, I am surprised. Με, εντυπωσιάζει ότι εδώ σε μια ακρόαση που ασχολείται με ένα θέμα τόσο σημαντικό για κάθε άτομο υπάρχει μόνο ένας άνδρας, το κοινό, ανάμεσά μας. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί άνδρες που έχουν αληθινό ενδιαφέρον για να ικανοποιήσουν και να αναγνωρίσουν πλήρως τα δικαιώματα των γυναικών. Η γυναίκα μου και εγώ έχουμε τρεις γιους και τρεις ε, γυναίκες. Και η γυναίκα μου μου είχε πει τη δεκαετία του 20, Μάριο, πρόσεχε πώς ε, συμπεριφέρεσαι προς τις κόρες μας, γιατί ανάλογα με τη συμπεριφορά σου θα αποδεχτούν τη συμπεριφορά άλλων αντρών στη ζωή τους, των συναδέλφων, συμμαθητών τους ή των μελλοντικών συζύγων τους. Και πραγματικά αυτό το έβαλα βαθιά στην καρδιά μου. Ποτέ δεν χτύπησα καμία από τις ε, κόρες μας, ούτε και τους γιους μας άλλωστε. Ποτέ δεν τις προσέβαλα, ποτέ δεν ύψα τη φωνή ποτέ δεν τις γελιοποίησα, ποτέ δεν τις ηρωνεύτηκα και τώρα έχουν και τον σεβασμό των συζύγων τους και οι τρεις μαζί έχουν 11 παιδιά συνολικά και νομίζω ότι θα έπρεπε στο πλαίσιο της εργασίας μας να προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε περισσότερους άνδρες όσον αφορά τέτοια θέματα που αφορούν τα αίτια αλλά και τις επιπτώσεις της φτώχειας, νομίζω ότι θα έπρεπε να προσθέσουμε επίσης την τοξικομανία, τον αλκοολισμό, την έλλειψη αυτοσεβασμού και την ε, ελευθεριάζουσα συμπεριφορά σεξουαλικά. Όσον αφορά τις ε, γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες τους τις παιδιά, ε, για κάθε τέτοια γυναίκα, φτωχή και μόνη και εγκαταλειμμένη, αντιστοιχεί επίσης υπάρχει ένας άντρας ε, μόνος και φτωχός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις απόψεις. Θα μπορούσα να έχω μια παρουσίαση εγώ λέγομαι Μάριο Ζέφκοβιτ. είμαι από το Ζάγκρεπ της Κροατίας και μαζί με τη γυναίκα μου είμαστε διευθυντές ενός οικογενειακού κέντρου ε, ε, κέντρου οικογενειακού προγραμματισμού στο Ζάγκρεπ που εξασφαλίζει μια πετυχημένη οικογενειακή ζωή. Πολύ σας ευχαριστούμε. Νομίζω λοιπόν ότι σίγουρα θα έχουμε κάποια σχόλια εδώ από το πάνελ Απλώς να πω η ίδια, έχουμε μελέτες που δείχνουν ότι οι κόρες οι οποίες έχουν τη σωστή αντιμετώπιση από τους πατέρες τους, αποδείχθηκαν σε συνέχεια δυνατές και ικανές στην κοινωνική ζωή. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να κάνει κάτι επιπλέον πριν να δώσω το λόγο στο πάνελ. Δεν βλέπω κάτι. Καλώς. Ε, ξεκινάμε με, τα, με τις σχόλια απαντήσεις από το πάνελ. Πριν να δώσουμε το λόγο στην κυρία Πλάμ. Παρακαλώ λοιπόν, ποιος θέλει να θα πάρει πρώτο το λόγο. Η κυρία. Ναι, καταρχήν θα ήθελα να τονίσω το πόσο τα δικά μας ε, μέλη υπολογίζουν στη δική σας ε, δουλειά ε, των βουλευτών για τη βελτίωση αυτών των θεμάτων. Έχουμε πολλά δίκτυα αυτή τη στιγμή και υποστηρίζουν τα αιτήματά μας όσον αφορά, για παράδειγμα, τη βελτίωση ζωής των γυναικών. φροντίζουν για τις γυναίκες αυτές, γιατί είναι ένα θέμα θεμελιωδών δικαιωμάτων και θεωρούν ότι δεν θα πρέπει 15 χρόνια μετά να συνεχίσουμε να, έχουμε, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Παρ' όλα αυτά η συζήτηση αυτή συνεχίζεται και θα συνεχίσει για πολλά χρόνια όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, υπολογίζουμε στη δική σας εισφορά και ε, μιλήσαμε για τη λεγόμενη εξατομίκευση των δικαιωμάτων. Ε, ναι, συμφωνώ, αλλά θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες συνήθως έχουν μόνο την σύνταξή τους. Ε, θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε τους ώστε να υπάρχουν κάποιοι μεταβατικοί μηχανισμοί να έχουν επαρκή συνταξιοδοτικά δικαιώματα οι γυναίκες αυτές. Επίσης, εκτιμώ το γεγονός ότι η Κομισιόν αναφέρθηκε στη βελτίωση της ε, φροντίδας για τα παιδιά. Νομίζω ότι η κατάσταση σε ορισμένες χώρες είναι ανισχυτική σε αυτό το τομέα και οι τοπικές αρχές πολλές φορές ε, αγωνίζονται γιατί έχουν πολύ περιορισμένους πόρους για την ε, φροντίδα των παιδιών ε, και περικόπτονται συνέχεια. Αυτό αφορά γυναίκες που εργάζονται αλλά και γυναίκες που ζουν περισσότερο από τους άνδρες και χρειάζονται συνεχή φροντίδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ με την κυρία Πάρενς. Και πριν να δώσω το λόγο, ή μάλλον καλύτερα να το κάνω τώρα, να δώσω το λόγο στον κύριο Κόχο. I agree very much. Δύο σχόλια. Συμφωνώ με αυτά που μας είπε η κυρία Φιγκουερέιδο. Θα μπορούσαμε να πούμε ίσως ότι το καλύτερο αποτέλεσμα του έτους κατά της φτώχειας είναι το ο στόχος για τη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη στρατηγική του 2020. Δεν συνδέονται, αλλά χωρίς το έτος κατά της φτώχειας θα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα να κάνουμε κάτι και να συμπεριλάβουμε κάτι για τη φτώχεια στρατηγική του 2020. Και θα μπορούσα ίσως να το πω και πιο ομά στη χώρα μου, τα προγράμματα που έχουμε εκεί τα κυβερνητικά δεν εμπεριέχουν σοβαρούς στόχους καταπολέμησης της φτώχειας μέχρι τώρα. Δεν έχουν θέσει σοβαρούς στόχους. Και αυτή η στρατηγική σπρώχνει το κοινοβούλια μας, τις κυβερνήσεις μας να κάνουν κάτι. τόσο αφορά και τους αριθμητικούς στόχους. Δύσκολο να εργαστεί κανείς με αυτά. Ανησυχώ λοιπόν λίγο. Εφαρμόζουμε εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα βιαστικά. Και αυτή η βιασύνη ίσως σημαίνει ότι δεν έχουν εξεταστεί σε αρκετό βάθος. Ότι ίσως δεν θα ανταποκριθούν ε, στους στόχους του 2020. Εγώ θα ήλπιζα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, πώς να το πω, θα έπρεπε να έχουν στη διάθεσή τους χρόνο για καλύτερη διαμόρφωση πολιτικής. Να μην βιαζονται υπερβολικά. και να χρειάζεται αυτό που θα θεσπίσουν πάρα πολύ γρήγορα μια ριζική μεταρρύθμιση σε μερικά χρόνια. Αυτά. Ευχαριστώ. Και θα περάσουμε στην κυρία Βασιλιάδου τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην επιδείνωση της καταστάσεως όσον αφορά τις γυναίκες που ζουν στη φτώχεια. Συμφωνούμε μαζί σας ήταν ένα από τα πορίσματα, όχι μόνο αυτά που αναφέρατε, και στην έκθεση που συντάξαμε την Oxfam είδαμε ότι η οικονομική κρίση αύξησε το ποσοστό των γυναικών στη φτώχεια και σημαντικά. Θα ήταν πολύ καλό να το εξετάσετε και αυτό. Όσον αφορά τις κατακαιρματισμένες πολιτικές εν συγκρίση με τις ολιστικές, αυτό προσπαθούμε να πούμε διότι παρακολουθώντας εξουσύνεγγες τις πολιτικές είδαμε ότι τα αποτελέσματα των πολιτικών είναι κατακαιρματισμένα. Και αυτό αφορά και τους στόχους του 2020 για τη φτώχεια ή για την απασχόληση των γυναικών και 75% απασχόληση των γυναικών. Τα αριθμητικά στοιχεία ίσως λένε ελάχιστα πράγματα να οδηγούν σε βιαστικά αποτελέσματα εκτός αν είναι σαφείς οι στόχοι που ακολουθούνται με σαφείς δείκτες και ορισμούς. Αλλιώς διατρέχουμε περισσότερους κινδύνους. Αυτά που είπε η Αν Σοφή ήταν σωστά. Χαιρόμαστε που λάβατε υπόψη τη φροντίδα των παιδιών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ηλικιωμένου και τα ατομικά εξατομικευμένα δικαιώματα. Να δούμε πού θα φτάσει αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνετε και ελπίζουμε να συνεργαστούμε. Ε, όσον αφορά τα όσα είπε, αναφέρθηκαν για τη συμμετοχή των ανδρών. Άκρος ευπρόσδεκτο από την οργάνωσή μας αυτό. Θα ήταν υπέροχο να είχαμε άντρες στην αίθουσα. Περιγράψατε ένα καλό παράδειγμα. Πως κάποιοι άντρες και γυναίκες μεγαλώνουν τα παιδιά τους με επικοδομητικό τρόπο μεγαλώντας μαθαίνουμε ότι η οικογένεια καμιά φορά είναι ασφαλής παράδεισος, καμιά φορά δεν είναι. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα μόνο εκεί. Υπάρχει διαφορά των αμοιβών, νομικές αβεβαιότητες, διάκριση νομική, πολλές άλλες αβεβαιότητες και δεν είμαστε ασφαλείς από όλα αυτά. Θα πρέπει όλα αυτά τα προβλήματα να εξαλειφθούν. Και ευχαριστώ που με καλέσατε να έρθω εδώ. Yes, please. Έχετε τον λόγο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μία διευκρίνηση. Το αίτημα για την εξατομίκευση των δικαιωμάτων ε, το θέτω προσωπικά σαν κάποιος που εργάστηκα πάνω στο θέμα της ισότητας των φίλων για αρκετά χρόνια και είναι μια έκκληση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το συμπεριλάβει ως αίτημα στην έκθεσή του δεν ε, προβάλλεται μέχρι στιγμής στην ε, στρατηγική των προσεχών ετών για την ισότητα των φύλων. Αλλά είναι μια έκκληση που θα μπορούσε να εκπληρωθεί ενδεχομένω. Και αυτό το λέω γιατί δεν θα ήθελα να δημιουργηθούν τυχόν ε, παρανοήσεις εδώ από τα όσα είπα. Καλώς, ευχαριστώ. Σίγουρα υπάρχουν συναδέλφ, συναδέλφεις εδώ που θα πάρουν, θα δράξουν αυτές τις ευκαιρίες και αυτές τις προκλήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα θα δώσω το λόγο στην ε, εισηγήτριά μας, αρμόδια εισηγήτρια, την κυρία Ροβάνα Πλάμ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Doresc să mulțumesc foarte mult ε, tuturor celor care Καλώς ευχαριστώ ε, όλους όσοι λάβανε μέρος στις συζητήσεις και για τις προτάσεις που έχουν γίνει για να βρούμε κάποιες λύσεις. Ειλικρινά με τιμά το ότι είμαι εισηγήτρια και είμαι πεπισμένη ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε μια πολύ καλή ομάδα διότι ειλικρινά θεωρώ αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας που υπάρχει στη στρατηγική αν όντω θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να, να είναι ανταγωνίσιμη μια Ευρώπη η οποία είναι σωστή με όλους τους πολίτες, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι χρειάζονται ε, συγκεκριμένα μέτρα. Και εμείς εδώ πέρα, οι βουλευτές της Ευρώπης που εκπροσωπούμε 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, πραγματικά εμείς θα πρέπει να έχουμε μια πιο ας πούμε ρεαλιστική προσέγγιση. Θα ήθελα να πω ότι προς το παρόν εμείς θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Ιδιαίτερα δύσκολη. Κυρίως στο ανατολικό μέρος της Ευρώπης. Διότι ειλικρινά ε, η φτώχεια που πλήττει τις γυναίκες είναι ακόμα πιο έντονη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Να μην επαναλάβω τι, τώρα κάτι από ό,τι έχει ελεγχθεί για τη γεωγραφική διάσταση δηλαδή, αλλά να πω ότι υπάρχει το θέμα που έχει να κάνει με τα δύο φύλλα. Εμείς από την πλευρά μας θεωρούμε ότι όσον αφορά τον διάλογο, τον κοινωνικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, επίσης με αυτούς που εκπροσωπούν ε, άλλους οργανισμούς, θα πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα, ούτω ώστε οι πολίτες να βρουν τις καλύτερες λύσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή, την εκπρόσωπη της Επιτροπής που ήρθε εδώ, διότι όντως η Επιτροπή θα πρέπει να μας δώσει μια βοήθεια θεσμική θα έλεγα. Μια δυνατή ε, υποστήριξη για να πετύχουμε, αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Επίσης, να πω ότι θα λάβω υπόψη όλα όσα ελέγχθησαν στι συζητήσεις, τόσο τις ε, κριτικές προσεγγίσεις όσο και τις προτάσεις και να πω σαν ε, μέλος στην Επιτροπή Απασχόλησης, εγώ άμεσα συνέβαλα σε, με κάποιες τροπολογίες για πάμε προς την σωστή κατεύθυνση όσον αφορά την απασχόληση. Γι' αυτό να πω θα ήθελα όμως να πω ότι δεν θα το πράξω αυτό μόνο, μόνοι, αλλά με όλους εδώ τους συναδόλφους, συναδέλφους, στην Επιτροπή και τους κοινωνικούς ε, ε, τέρους, καθώς και τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, να προσπαθήσαμε να πετύχουμε τους στόχους μας, να διασαφηνίσουμε τα θέματα, να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε την απασχόληση στην αγορά εργασίας, να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες. Επίσης, το θέμα του χάσματος όσον αφορά ε, στην, ε, στην μισοδοσία, που όλοι μιλάμε γι' αυτό. Μια εξαρτία, να βρούμε συγκεκριμένα μέτρα, ούτως ώστε να το αντιμετωπίσουμε και αυτό το πρόβλημα. Επίσης υπάρχει το θέμα για τις ε, συντάξεις, η πράσινη βίβλος. Εμείς στην ομάδα μου, οι σοσιαλιστές, έχουμε ασχοληθεί πολύ με αυτό το θέμα της πράσινης βίβλου της Επιτροπής. Οι χώρες μέλη έχουν εδώ πέρα να κάνουν πάλι με μια στρατηγική όσον αφορά τα συστήματα συντάξεως. Στη Ρουμανία φέρει πίν. Εμείς έχουμε μια κατάσταση όπου βλέπουμε πολλές γυναίκες άμα δει κανείς ότι θα 65 ετών σαν όριο συνταξιοδότης τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες μετά το πέρασμα στη συνταξιοδότηση, τότε οι γυναίκες ε, σε σχέση με το προσδόκιμο ζωής οδηγεί δηλαδή σε ε, ακόμα μισή χρόνια. Στη Ρουμανία δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι ε, αυτό το θέμα δεν αντιμετωπίστηκε σωστά και είναι κάτι το οποίο επίσης θα θίξουμε. Στι χώρε όσον αφορά στο ανατολικό μέρος της Ευρώπης, σκέφτομαι την Ρουμανία, τη Βουλγαρία, που περνάνε μια μεγάλη κρίση όσον αφορά τις μειονότητε, εθνικές ε, Φέρει Φερρυπίν υπάρχει ο προβληματισμός για τους ε, Ρώμα, που πρέπει να προχωρήσει. Μετά έχουμε το θέμα της αγοράς εργασία, ενό συστήματο για τι συντάξει το οποίο θα πρέπει να είναι βιώσιμο, ο συνδυασμός ε, ιδιωτική οικογενειακής ζωής και επαγγελματική, ε, τη φροντίδα των παιδιών και για το πώς μπορούμε να έχουμε μια κοινωνική ασφάλιση η οποία είναι βιώσιμη, ε, η φροντίδα των ηλικιωμένων. Είναι όλα αυτά θέματα τα οποία θίγουμε. Είναι υπηρεσίε όλα αυτά. Επίσης έχουμε το θέμα τι γίνεται με τις οικογένειε, όπου μόνο ένας συμβάλλει οικονομικά για την συντήρηση τη οικογένειας. Ε, επίσης οι οικογένειες οι οποίες έχουν κάποια μεγάλα προβλήματα όπου φέρνει να έχουμε γυναίκες που έχουν προβλήματα κινητικά, παιδιά με ανάλογα προβλήματα, γυναίκες μετανάστριες. Όλα αυτά τα θέματα θα είναι μέρος της ε, έκθεσης. Επίσης, οι επιπτώσεις ε, της φτώχειας, ε, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η βία, η εμπορία λευκής σαρκός. Επίσης, όπως ανέφερε και η κυρία υπάρχει το θέμα του ελάχιστου εισοδήματος. είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα. Και ελπίζω ειλικρινά να, να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια πολιτική απόφαση. Μια καλή ιδέα επίσης είναι να δούμε τα δικαιώματα όσον αφορά την, ε, ας αφορούν την ε, εξατομικεμένη ε, ασφάλιση. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συγκεκριμένα, συγκεκριμένες προτάσεις αλλά για να πετύχουμε, αν όντω θέλουμε να πετύχουμε, χρειαζόμαστε και τους ανάλογους πόρους. Γι' αυτό, επαναλαμβάνω, στην Επιτροπή, βοηθήστε μας, υποστήριξτε στη, αυτήν εδώ την έκθεση ε, και να εξασφαλιστούν ε, με υπολογισμό Τα οποία κονδύλια θα πρέπει να ε, σε αυτούς εδώ τους στόχους. Αν η Επιτροπή ε, δει στον προπολογισμό να υπάρχουν κατάλληλοι πόροι για θέματα ισότητας, τότε ειλικρινά μπορούμε να πούμε ότι ίσως να πετύχουμε. Τώρα κοιτάξτε, ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι σε σχέση με αυτά που ελέγχθησαν. Ε, θέλω να υπογραμμίσω την οδηγία που αφορά την προστασία την εργασία, ε, στο χώρο εργασίας η Επιτροπή Απασχόλησης είναι υπεύθυνη που έχει να κάνει με, αυτό το θέμα και με την ε, γονική άδεια και τις επιπτώσεις που μπορεί να, υπάρχει, να υπάρχουν σε μια γυναίκα. Δηλαδή η γυναίκα να μην πλήτεται στο, από διάφορες επιπτώσεις στο χώρο εργασίας. Η γυναίκα φέρει πίνη, για ένα, ένα παιδί. Ε, χάνει ένα μεγάλο μέρος από το μισό της. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Δηλαδή κάθε διαφορά που υπάρχει οδηγεί σε, στο ότι πλήττεται η γυναίκα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε μια πολιτική η οποία θα πρέπει να είναι αποτελεσματική όσον αφορά την ισότητα και για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ε, ε, βλέπουμε αυτό το θέμα που συζητάμε πολύ, το mainstreaming. Αυτό πρέπει να το δούμε σε όλε τι πολιτικές. Και τέλος, να κλείσω λέγοντας, ε, εμείς θέλουμε να δουλέψουμε από κοινού. Και είμαστε ε, θετικοί. Άσχετο αν τώρα μιλάμε σαν, ε, όταν, έχουμε να μιλάμε σαν Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, κοινωνική εταίροι, θα είμαστε θετικοί, θα ελπίζω να έχουμε μια ε, επιτυχία. Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις προτάσεις, να λειτουργήσουμε σαν μια ομάδα και πιστεύω θα υπάρξει μια, θα λέγαμε, εταιρική σχέση, μια σωστή συνεργασία με όλες τους όσοι συνεργάζονται σε αυτήν μας εδώ την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Πλάμ, λέει πρόεδρος. Είμαι πεπισμένη ότι θα έχουμε σωστή συνεργασία και θα έχουμε ε, πρόοδο στους στόχους μας υπάρχει ε, ε, η δέσμευση όλων. Ε, εντάξει, είχαμε μια μέρα η οποία, ε, στην οποία αντιμετωπίσαμε και κάποια τεχνικά προβλήματα, το ξεπεράσαμε. να καταλήξω ευχαριστώντας εδώ τα μέλη στο Προεδρείο, τους καλεσμένους μας, τις καλεσμένους, τις καλεσμένες στο πάνελ, να, να εκφράσω τις ευχαρισίες μου στην εκπρόσωπο της Επιτροπής, στις συναδέλφους και συναδέλφους, όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτήν εδώ την ακρόαση επίσης στη γραμματεία. Και φυσικά, τέλος, αλλά εξίσου σημαντική, η συμβολή της Γερμηνίας. Σας ευχαριστώ όλους. Καλό σας βράδυ.